να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ε, συνεδρίαση μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Ε, σας ε, καλωσορίζω όλους. Θέλω να σας ευχηθώ και καλή χρονιά και ελπίζω όλοι να έχουν ξαναγεμίσει τις μπαταρίες τους κατά διάρκεια των θερινών διακοπών. διότι ξεκινάει πάλι η δουλειά, έχουμε νέα Προεδρία του Συμβουλίου και έχουμε πολλά θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Πολύ, πολύ δουλειά μας περιμένει. Εύχομαι πάντως ε, κυρίως μια καλή ε, χρονιά και με υγεία. Το σημείο 25 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση Ούλμερ. θα αναβληθεί για τις 19 ε, Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η μόνη τροποποίηση. Αν δεν υπάρχει άλλη αντίρρηση, εκρίνεται η μέρη σε διάταξη ως έχει. Έχουμε όλες ε, τις γλώσσες ε, στην διερμηνία και και ε, μαλτέζικα, κροατικά ε, και βλέπω νομίζω να τις χρησιμοποιήσουμε. Από τις 5 ε, μέχρι τις 6 θα έχουμε προσκεκλημένους τον δήμαρχο της περιοχής Ρουρ, ο οποίος εκατό με δική μου πρόσκληση θα συμμετάσχει στην σημερινή συνεδρίαση. Δεν υπάρχει διαμηνία στα αγγλικά, παρακαλούμε μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωραία. Ωραία, όλα καλά. Επαναλαμβάνω, από τις 5 μέχρι τις 6 θα έρθει ο, ε, ο δήμαρχος ε, της περιοχής Ρουρ ε, και θα συμμετάσχει στην συνεδρίασή μας. Άλλωστε έχουμε αρκετές θέσεις στη διάθεσή μας. Επίσης ε, θα έχουμε ομάδα του BBC που θα κάνει ε, που ε, θα, θα κάνει ηχογράφηση ε, και επίσης ε, έχουμε μία επιπλέον εκπαιδευτική συνάντηση. Έχουμε εισάγει τώρα το σύστημα των ε, συνεδριάσεων χωρίς χαρτί, ηλεκτρονικά δουλεύουμε. Καλό λοιπόν τους ε, συναδέλφους ε, σήμερα και αύριο από τις 2 έως τις 2.30 να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις ηλεκτρονικές επιτροπές ή κομίτη. Πέμπτη ανακοίνωση. Έχουμε στείλει αντιπροσωπεία στην Κροατία. Η έκθεση της αντιπροσωπείας υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΝΒΗ. Όποιος θέλει πληροφορίες μπορεί να προσφύγει εκεί. Φτάνουμε στην έγκριση των πρακτικών. Ε, είχαμε ε, την ακρόαση στις, ε, του, του Μπορζ 12 Νοεμβρίου και τη συνεδρία στις 13 Νοεμβρίου. Ωραία και περνάμε τώρα στον ε, προσκεκλημένο μας. Ε, ξεκίνησε η Προεδρία της Ιρλανδίας και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Γεωργίας, Διατροφής και Θαλασσίων Θεμάτων, ε, τον Υπουργό Σάιμον Κόβενι. Πολύ δουλειά σας περιμένει η γεωργική μεταρρύθμιση που αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων, η μεταρρύθμιση στην Αλία και άλλα πράγματα. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά για το Κοινοβούλιο, για τους εισηγητές, ε, αλλά και για ε, την Προεδρία της Ιρλανδίας. Θέλουμε λοιπόν ε, σήμερα να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας, να ακούσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας Ως ε, ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, έχουμε υιοθετήσει γνωμοδότηση για την αλληλεία αλλά και για τη μεταρρύθμιση της, γεωργίας, της γεωργικής πολιτικής. θα θέλαμε λοιπόν να δούμε να λαμβάνονται υπόψη οι γνωμοδοτήσεις μας στα θέματα αυτά. αλλά ε, σύντομα θα έχουμε τη ε, δυνατότητα να συνομιλήσουμε και κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much, uh, Chair. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να κάνω αυτή την παρουσίαση και βεβαίως να κάνουμε και μετά ένα κύκλο ερωταπαντήσεων με την Επιτροπή. Σας γνωρίζω το γεγονό, ε, καθώ έχω υπάρξει Ευρωβουλευτή στο παρελθόν, τη σημασία που έχει αυτή η Επιτροπή. Είναι μία από τι πλέον βεβαρημένε με εργασίε Επιτροπή του Κοινοβουλίου και τα καθήκοντά σα αφορούν ευρύτατα τους τομείς από το περιβάλλον, τη γεωργία, την αλλαγή του κλίματος και τόσα πολλά α, επιμέρους θέματα όπως είναι η ευημερία των ζώων, η επισήμανση κτλ. Γνωρίζω λοιπόν ότι και σήμερα έχετε επιβαρημένη Μυρίστα διατάξη. Τρει ε, Ιρλανδοί υπουργοί σα κάνουν μια παρουσίαση. Ο Υπουργό Γεωργία, Υπουργό Περιβάλλοντο και ο Υπουργό Υγεία θα σα κάνουν μια παρουσίαση. Οπότε είναι καλό να ξεκινήσουμε το πρωί με τα γεωργικά ζητήματα. Θέλω να επισημάνω πάντως ότι το επόμενο εξάμεινο εμείς έχουμε υιοθετήσει μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα, την οποία παρουσιάσω σε λίγο, σε ό,τι αφορά τη γεωργία και την αλληλεία και τα συναφή ζητήματα. Διότι η, Συλλογική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, συλλογικά, στην προσπάθεια να οριστικοποιήσει την κοινή αγροτική πολιτική κοινή λιχτική εποχή με ένα νέο μηχανισμό λήψη αποφάσεων βάση Λισαβόνα είναι κάτι πραγματικά καινούριο. Δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και θα πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνει με τα περισσότερα κράτη-μέλη που είχαμε ποτέ. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη πολιτική πρόκληση και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και σε ό,τι αφορά την διαδικασία τη απόφαση, όπω και τα επιμέρου θέματα. Θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε ε, σε ένα πρωτοφανέ χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αποφάσεων, η διαδικασία του τριμερούς διαλόγου και η συναπόφαση ελπίζουμε και για τους δύο μεγάλους φακέλους, για την κοινή αγροτική πολιτική και η κοινή ληφτική πολιτική, να ολοκληρωθούν μέσα στην ε, Ιρλανδική Προεδρία. Ένας από τους λόγους τους οποίους επιμένει αυτή η Προεδρία και γι' αυτό ορίσαμε φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ε, η εναλλακτική λύση ήταν πολύ επικίνδυνη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, α, να περιμένουμε ουσιαστικά στο τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου σας για να κλείσουμε τους φακέλους. Για πρακτικούς αλλά και πολιτικούς σε κάποιες περιπτώσεις λόγους θα ήταν προβληματικό αυτό, γιατί υπάρχουν α, διάφορες εκλογές που εκκρεμούν, μεταξύ αυτών και ευρωεκλογέ του χρόνου. Ε, δράτω με ευκαιρία την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες τη Προεδρίας μας, ιδίως σε ό,τι αφορά τα θέματα που αφορούν την δική σας ε, Επιτροπή. Θα εστιάσω συγκεκριμένα στην, ε, στις για την ε, κοινή ελευθερική πολιτική που θα πρωταγωνιστήσουν το επόμενο διάστημα, αλλά και γενικότερα ποιες είναι οι προτεραιότητες της Προεδρίας μας και να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα αυτό και για τις άλλες ομαδικές προτάσεις που είναι στο τραπέζι ή που τι τις περιμένουμε. Λίγα λόγια για τους γενικότερους πολιτικούς στόχους της Προεδρίας. Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε σε τρεις λέξεις, ε, αν θέλει το σλόγγαν τη Προεδρία. σταθερότητα, θέσει εργασία και ανάπτυξη. Θέλουμε να βελτιώσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Άρα λοιπόν οι τομιακές ε, πολιτικές μας προτεραιότητες έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια νέα βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια στρατηγικής Ευρώπη 2020. Τώρα να ε, πάω σε θέματα γεωργίας και αλληλεία. Οι συζητήσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα κυριαρχηθούν από τι διαπραγματεύσει για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική και κοινή αλληλευτική πολιτική. Και δύο πακέτα πολύ σημαντικά για να διαμορφώσουμε τη μελλοντική δομή α, του τομέα γεωργία και τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχο είναι να έχουμε μια συνολική πολιτική συμφωνία και για τα δύο πακέτα ω τα τέλη του Ιουνίου 2013 και θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο. Σε ό,τι αφορά άλλους φακέλους ε, που έχουμε αναλάβει, η Κομισιόν προτίθεται να δημοσιεύσει ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων για την υγεία των οζών και των φυτών, επίσημη, επίσημους ελέγχους και τους σπόρους, το δεύτερο τρίμηνο του 2013 κάτι που περιμέναμε πέρυσι ουσιαστικά, αλλά τελικά θα έρθει γύρω στο Μάρτι. Μια πολύ σημαντική δέσμευση δημοτικών προτάσεων ώστε να έχουμε σε ενοποιημένα κείμενα, αλλά και εξυγχρονίζοντας ταυτόχρονα, τον πυρήνα της, ε, των αναμονισμένων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ε, ζώων και των φυτών. Η Ελληνική Προεδρία θα ηγηθεί των συζητήσεων στο Συμβούλιο, ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή πρόοδο έως τον Ιούνιο. Ένα στοιχείο αυτού του πακέτου είναι η πρόταση κανονισμού για τα τρόφιμα και τις οτροφές και τις δαπάνες συγκεκριμένα αναμένεται να δημοσιευτεί το Φλεβάρι και η Ιρλανδία θα θέσει ως βασική προτεραιότητα τις συζητήσει, ώστε να επιτύχουμε πρόοδο έως την ημερομηνία στόχο για φέτος που είναι η 31 Δεκεμβρίου 2013 να περάσει αυτή η νομοθεσία. Δεν θα αρνηθώ ότι έχουμε πολλές διαδικαστικές ε, προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αυτό το πακέτο. Το στοιχείο δαπανών συνδέεται με το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, το οποίο θα πρέπει να θέσει σε ισχύ από 1η 2014. Η Ελληνική Προεδρία είναι έτοιμη έτοιμη στο πλευρό του Συμβουλίου να καταβάλει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία και με την Επιτροπή προς την ίδια κατεύθυνση επίσης. Σε ό,τι θέλω την πρόταση για το μέλη. Κάποιοι στην Επιτροπή σας ε, ξέρουν ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η πρόταση αυτή α, ξεκίνησε να εξετάζεται από την Ελληνική Προεδρία με την πρώτη τεχνική εξέταση τη πρόταση να γίνεται σε επίπεδο της εργασίας 18 Γενάρη. Πρόταση αυτή έχει στόχο να διευκρινίσει το καθεστώ ε, τη γύρης ω φυσικό στατικό ε, του μελιού και ε, κάτι διαφορετικό δηλαδή από το υλικό και αυτό απαιτεί κάποια θέματα ευθυγράμμιση. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή σα έχει ξεκινήσει την εξέταση τη πρόταση και προσβλέπουμε στο αποτέλεσμα τη συζήτηση που θα γίνει και εδώ στην Επιτροπή σα αύριο. Θεωρούμε ότι μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση με το Κοινοβούλιο είναι κάτι εφικτό έως τα τέλη του Ιούνιου 2013. Περιμένω να συνεργαστούμε από αυτού μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι έχουμε σημαντικές αποκλήσεις ανάμεσα στο Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ε, τα άπαντα ε, για το πρωινό το breakfast omnibus όπως ε, λέμε. είναι κάτι που η Επιτροπή σα και ο Πρόεδρος σας γνωρίζετε πολύ καλά. Το σχέδιο κοινωνισμού για τις λεγόμενες οδηγίες πρωινού συνδέεται με την ε, εξουσία ευθυγράμμισης που δίνεται στην Κομισιόν από τη Συνήθεια Λαβόνε. Αφορά πέντε συγκεκριμένα προϊόντα και σχετικές οδηγίες που είναι η σοκολάτα, ο καφέ, η ζάχαρη, οι μαρμελάδες ε, και το κομμένο γάλα. Γενική ε, προσέγγιση στο Συμβούλιο έχει συμφωνηθεί και από ό,τι γνωρίζω η θέση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για αυτό το φάκελο είναι πολύ κοντά, ποτέ δεν ταυτίζονται, το γνωρίζετε αυτό. Άρα λοιπόν η Ελληνική Προεδρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσει στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν από την αρχή του Μαρτίου. Δηλαδή, όταν υφηθεί η Επιτροπή σα το σχέδιο έκθεση, που, αν γνωρίζω καλά, προβλέπεται να υφηθεί στις 20 Φεβρουαρίου. Σε ό,τι αφορά ε, το, την πρόταση για την μη εμπορική ε, διακίνηση ε, των ζώων είναι ένας φάκελος που ξεκίνησε να εξετάζεται από την Κυπριακή Προεδρία και εμείς θα κάνουμε τον τρίτο γύρο τριμερούς διαλόγου για αυτό το θέμα. Θα συζητήσουμε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση βοηδών και την εθελοντική σήμανση ε, των βοηδών. Και για τις δύο προτάσεις είναι φιλόδοξη η προσέγγιση μας και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση αν υπάρχει συμφωνία και με το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη δασοκομεία, η Επιτροπή σας έχει ξεκάθαρες θέσεις θέσεις επί του θέματος. Διαπραγματεύσεις για ε, ένα LBA ε, για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινηστεί και δύο τελευταίες συζητήσεις προβλέπεται να γίνουν στο πρώτο εξάμεινο 13. Ο συνολικός στόχος είναι επέκταση συμφωνία που θα αποτελέσει ορόσημο για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στην Ευρώπη. Η Λονδική Προεδρία θα κάνει κάθε προσπάθεια για να διευκολύνει την πρόοδο προ αυτή τη συμφωνία και θέλω να προσθέσω ότι αναμένεται ότι και η Κομισιόν θα δημοσιεύσει μια στρατηγική για τη δασοκομεία του επόμενου μήνε που θα θέσει το πλαίσιο τη συζήτηση για τη μελλοντική διαχείριση του δικτύου δασών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι κλείνω την παρουσίασή μου για αυτά τα ζητήματα. Θέλω όμω πολύ καλό για παραπάνω για του δύο βασικού φακέλου που ειλικρινά πρέπει να ομολογήσω θα κυριαρχήσουν ε, στις σκέψεις μου και τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε στο επόμενο εξάμεινο στο Συμβούλιο. Πρώτα απ' όλα, μεταρρύθμιση κοινή ελληνική πολιτική. Χθε είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με την ε, Επιτροπή Αλληλείας για το φάκελο αυτό. Η Ιρλανδική Προεδρία έχει ως πρώτη προτεραιότητα να επιτύχει πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το περιεχόμενο αυτού του πακέτου μεταρρύθμισης κοινή ελευτικής πολιτική. Για κάθε κανονισμό μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία είτε στην πρώτη ανάγνωση ή ε, νωρί στη δεύτερη ανάγνωση. Όμω αυτό απαιτεί δέσμευση από όλε τι πλευρέ, Συμβούλιο, Κομισιόν ε, και βεβαίω και από τη δική σα πλευρά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ελληνική Προεδρία είναι έτοιμη να ξεκινήσει διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται νωρίτερα, ώστε να διευκολύνουμε την επίτευξη πολιτική συμφωνία ανάμεσα νομοθέτε. Το πακέτο μεταρρύθμισης απαιτεί και τα δύο όργανα να εργαστούν γρήγορα χωρίς όμως να πιέσουν τι αποφάσεις. Πρέπει όμως να δουλέψουμε γρήγορα και σε στενή αγαστή συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι αφορά την ρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική, το έχω ξαναπεί. Στόχο Ιρλανδία είναι να διασφαλίσει πολιτική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα έω το τέλη του Ιούνιου να μην ξεχνάμε ότι συζητούμε αυτή τη μεταρρύνση της ΚΑΠ εδώ και τέσσερα χρόνια. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να προχωρήσουμε και από τις συζητήσεις και τα λόγια να περάσουμε σε συγκεκριμένε δράσεις. Αυτό προσπαθήσει να κάνει η Προεδρία. Γνωρίζω απόλυτα ότι είναι πολύ φιλόδοξο αυτός ο στόχος ότι θα απαιτήσει εντατικέ εργασίε και μεγάλου συμβασμού από όλε τι πλευρέ, αλλά βασικά να συμβούν τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει συμφωνία για το πολιτισμο οικονομικό πλαίσιο όσο γίνεται νωρίτερα μέσα στο 2013. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πιο αισιόδοξοι ότι μπορεί να συμβεί στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο Κορυφή των Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων. είναι όλο και πιο πολλέ οι ελπίδε που μπορεί να υπάρξει συμφωνία τότε. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει γρήγορη πρόοδο στα εκκρεμή τεχνικά και πολιτικά ζητήματα ώστε να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου το στομότερο δυνατόν. Τα εκκρεμή ζητήματα έω τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολα για τι διαπραγματεύσει, όμω ελπίζουμε ότι θα κλείσουμε και θα καταλήξουμε στη θέση του Συμβουλίου έω το ορεινό Συμβούλιο, το Συμβούλιο του Μαρτίου αυτή τη προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την πραγματική μα θέση ε, για τα βασικά θέματα τη ε, μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ στο Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Και αυτό λειτουργεί παράλληλα με τι εργασίε του Κοινοβουλίου. Όταν και εσεί δηλαδή θα ολοκληρώνετε τη δική σα θέση στην Ολομέλεια του Μαρτίου για την ΚΑΠ. Και ε, ήδη σήμερα βλέπουμε ότι στην Επιτροπή Γεωργίας υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι ψηφοφοριών για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ξέρω ότι και η δική σας Επιτροπή έχει μια σειρά γνωμοδοτήσεων που συνδέονται με την ίδια διαδικασία. Αν η Ελληνική Προεδρία καταφέρει να οριστικοποιήσει την διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου έω το Συμβούλιο του Μαρτίου, τότε κατά τα όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν, θα πρέπει γρήγορα να ξεκινήσουν τη διαδικασία τριμερού διαλόγου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόφασης ω τα τέλη του Ιούνιου. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Η ορνή είναι θετική αυτή τη στιγμή. ότι Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιτύχει συμφωνία για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως είπα και πριν, ελπίζουμε ότι η συμφωνία θα είναι τέτοια ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να δώσει γρήγορα τη συνένεσή του. Θα το δούμε βεβαίω αυτό. Τούτο λεχθέντος, η πραγματικότητα είναι ότι η συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, δεν είναι απόλυτα στον έλεγχο αυτής της Προεδρίας ή της Επιτροπής σας. Οπότε θα πρέπει να στήσουμε προσοχή μα στου άλλου δύο όρου, άλλε δύο προποθέσει, τι οποίε μπορούμε να ελέγξουμε. Εγώ θα κάνω κάθε προσπάθεια να διασφαλίσω τη συμφωνία του Συμβουλίου για όλα τα κρεμμένα ζητήματα στο τέλη Μαρτίου. Δεν έχω ψευδεστήσει. Ε, είναι πολύ φιλόδοξοι αυτοί οι στόχοι και θα απαιτήσουν τεράστιε προσπάθειε και μεγάλου συμβιβασμού από όλε τι πλευρέ. Αλλά είναι ο μόνο τρόπο για να πετύχουμε του συνολικού στόχου και την πολιτική συμφωνία για αυτό το φάκελο του επόμενου μήνε. Αυτό θα απαιτήσει ε, μία συλλογική δέσμευση κατά εξαίρεση από όλα κατά τα τρία θεσμικά όργανα για να υπάρξει πολιτική συμφωνία μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Παρότι η Επιτροπή σας δεν έχει την κύρια ευθύνη για αυτό το φάκελο, γνωρίζω ότι έχει ενημερωθεί ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και ενδιαφέρεται σημαντικά και ε, λόγω των πτυχών του περιβάλλοντος και του προσυνείσματος ε, στο μεταρρύθμιση. Έχω καταγράψει προσεκτικά τις γνωμοδοτήσεις που έχετε συντάξει σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσει και τις προτάσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Όμως η δική μου δουλειά το επόμενο διάστημα ως προ... Ε, την Προεδρία του Συμβουλίου σε θέματα γεωργίας είναι διασφαλίσω μια ισορροπημένη συμφωνία αποδεκτή από όλους. Σε ό,τι αφορά το πρίπλοκα ζήτημα που ονομάζεται πρασίνισμα, greening, φαίνεται από την προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τον πυλώνα προσυνείσματος 1 ε, να υπάρχει μια ευρεία συμφωνία επί των προτάσεών της. Όμως υπάρχουν άλλα λεκτά ζητήματα που είναι τα ποσοστά ενεργοποίησης, ε, η ευελιξία και άλλα ζητήματα που άπτονται των γεωγραφικών και τοπογραφικών προϋποθέσεων. Φυσικά και θα ακολουθήσουμε την πρόοδο που επέτυχε η Εθνική και η Κυπριακή συγγνώμη, Προεδρία και συνεργασία με τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ελπίζουμε να επιτύχουμε τον επιθυμητό πόλου συμβασμό. Τέλος, θα ήθελα να πω πριν έλθω και κάνω αυτή την παρουσίαση, εδώ μπροστά σας διαβάζοντας την, αισθάνθηκα κάπως αμήχανα λόγω του όγκου και του μεγέθους αυτής της δουλειάς. Αν δείτε το εύρος και την ε, έκταση των διαφερόντων της Επιτροπής σας για θέματα που το του μου κατανοώ ότι μπορεί να θέσετε πάρα πολλές ερωτήσεις για πάρα πολλά ζητήματα και ελπίζω να είμαι προετοιμασμένος. Θέλω πάντως να σας δείξω ποια... ποιος είναι ο στόχος της ελληνικής προεδρίας για αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι αρμόδιοτά μου είναι κατά κύριο λόγο το πακέτο μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ τη πολιτικής, πολιτική, αλλά και τα λεπτά ζητήματα. Οπότε περιμένω τι ερωτήσει. Ευχαριστώ για τον χρόνο σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα έχουμε τώρα δύο γύρους ερωτήσεων. Ε, το γνωρίζετε και εσείς ε, ότι εδώ στο Κοινοβούλιο πρώτα έχουμε έναν γύρο με τις ερωτήσεις των συντονιστών και κατόπιν δίνουμε το λόγο στους ε, συναδέλφους. Καταρχήν να δώσω το λόγο στον Ρίχαρτ Σίμπερ, Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Προεδρεύοντα που ήρθατε εδώ για να μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα ε, της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ε, καταλαβαίνετε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το greening. Ήταν πολύ γενικές οι εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά μήπως ε, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες ε, σχετικά με τα συγκεκριμένα σχέδια σας ε, γνωρίζουμε την πρόταση ε, της Κομισιόν, το 30% του πρώτου πυλώνα θα πρέπει να αφορά το greening. Μπορείτε να δεχτείτε εσείς το ποσοστό αυτό ή ε, έχετε κάποια πιο ενδιαφέρουσα πρόταση. Γνωρίζετε τις ανησυχίες κρατών μελών που έχουν επενδύσει πολλά για μέτρα του πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Πώς θα υπολογιστούν λοιπόν τα μέτρα αυτά και οι πόροι που έχουν διατεθεί στον δεύτερο πυλώνα, ώστε αυτοί που ήδη έχουν προχωρήσει ένα βήμα πιο, πέρα να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση με την μεταρρύθμιση και τι γίνεται με τις ε, περιοχές ε, που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές περιοχές κλπ. Ε, Μπορούμε παράλληλα να ε, έχουμε αυτές τις δύο σειρές μέτρων ή ε, έχει ε, σκεφτεί κάτι άλλο ή το Συμβούλιο. Επίσης, τι γίνεται όσον αφορά την αγρανάπαυση. Η Κομισιόν έχει το ποσοστό του 10%. Πώς το βλέπετε εσείς και αναφερθήκατε και σε πρότυπα της Κομισιόν. Το Συμβούλιο τι λέει για αυτά. Επίσης, ε, μας περιμένουν ε, ε, τροπολογίες και ψηφοφορίες και από ό,τι κατάλαβα οι τροπολογίες είναι πολύ γραφειοκρατικές. Αυτό που επικρίνουμε ακριβώς το βρίσκουμε στις τροπολογίες. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να μειωθεί κάπως η ε, γραφειοκρατία και το θέμα της αλίας το αφήνω στους συναδέλφους ε, που ασχολούνται περισσότερο με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ ε, τον Ρίχαρτ Σέπερ, η Λίντα Μακέβαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα το πρωί. Προφανώ βλέπουμε ότι τα, οι βασικοί φάκελοι που, με του οποίου θα ασχοληθείτε θα είναι η αλληλεία και ε, η κοινή αγροτική πολιτική. μεταρρύθμιση αυτών των δύο και η Επιτροπή μα πάντα ασχολήθηκε με αυτά τα ζητήματα και θέλουμε να γίνει μια σωστή μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Ε, ξέρουμε ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντό για την Ελλαδική Προεδρία. Δεν, μπορούμε να έχουμε μέλλον ε, ε στον τομέα της ε, αλληλείας ε, εκτός και αν υπάρξει πραγματική δέσμευση από τους πολιτικού μας φορείς. Ε, έχουμε τώρα την πρόταση της Επιτροπής που είναι φιλόδοξη. Ελπίζω αυτή η πρόταση να μείνει ακέραια ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ίσως μπορείτε να μας πείτε τι συμβαίνει ακριβώς στο Συμβούλιο με τη μεταρρύθμιση τη ε, αλληλευτικής πολιτική. Ακούγεται ότι θέλουν τα κράτη-μέλη να αποδυναμωθεί σημαντικά η μεταρρύθμιση και να επιστρέψουμε στα παλιά, ότι ε, στα τέλη του Δεκεμβρίου, μέσα στη νύχτα, αποφασίσουμε να, διαπρα... διαπραγματευτούμε και να αποφασίσουμε για το μέλλον της αλληλευτικής πολιτικής. Τώρα, να θυμάστε ότι στην Ολομέλεια οι ψηφοφορίες μπορεί να μην είναι ίδιες ε, με την ε, ψηφοφορία στην Αγροτική Επιτροπή. Γιατί γίνονται πολλές, πολλοί συμβασμοί στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων. Επομένω, δεν αρκεί μόνο μια συμφωνία στην ε, Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων. Πρέπει στην Ολομέλεια να επιτευχθεί η συμφωνία. Ό,τι και αν γίνει με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ξέρουμε ότι πολλά από τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα κατευθυνθούν ε, στη γεωργία. Γι' αυτό είναι κάτι που μα απασχολεί. Τελευταίο ζήτημα, κάτι που βρίσκεται στην επικαιρότητα και στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο σιγά σιγά ακούγεται και σε άλλε χώρε το σκάνδαλο με τα ε, μπιφτέκια βοηδού ε, που έχουμε κρούσματα ε, και στην Ιρλανδία και στο Μενοβασίλειο και για το ε, κρέας αλόγου και στο χοιρινό. Κυρίως όμως για αυτά τα μπιφτέκια βοδινού ξέρετε τι συμβαίνει, πώς προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Και μετά ε, για την ε, επισήμανση ε, στα τρόφιμα. Το Κοινοβούλιο προσπάθησε να καταστήσει αυστηρότερο το νομικό πλαίσιο κατά την τελευταία αναθεώρηση και είπαμε ότι πρέπει να γίνεται εντοπισμός που μιλάμε για φρέσκο νοπό κρέας και που υπάρχει δευτερογενές προϊόν. υπήρξε συμβασμός με το Συμβούλιο ότι ουσιαστικά θα υπάρξει έκθεση από την Επιτροπή το 2014. Εξέτασα το τρέχον νομικό σύστημα και βλέπουμε ότι αυτά τα beef burgers που είναι 99% βοδινό πρέπει να λέμε ότι ποια είναι η χώρα προέλευσης. Αν όμως είναι μικρότερο το ποσοστό από 99% δεν, δεν χρειάζεται, αν υπάρχει δηλαδή ανάμειξη ε, κρέατος. Και έτσι είναι σαφές ότι οι μεγάλες αλυσίδες ε, πολυκαταστημάτων και σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται το προϊόν του και αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση το 2014 και μήπως ε, τώρα είναι αυτό κάτι που επανεξετάζεται από τους υπουργούς ε, στο Συμβούλιο. Ελπίζω οι συνάδελφοι από την άλλη πλευρά του Κοινοβουλίου να κατανοήσουν την σημασία της ε, κατάλληλης επισήμανσης τροφίμων. Φανταστείτε, κάποιοι από τους ε, ψηφοφόρους να δουν ότι ενώ για θρησκευτικού λόγους δεν ε, τρώνε χοιρινό κρέας, να συνειδητοποιήσουν ξαφνικά ότι τα προϊόντα που αγοράζουν εμπεριέχουν χοιρινό κρέας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λίντα Μακέβαν, ο Κρις Ευχαριστώ. Υπουργέ ο Πρωθυπουργό Κάμερον τη χώρα μου αυτή τη στιγμή κάνει μια ομιλία. Τι να κάνω, να ακούσω εκείνον ή εσά. Uh, Σα άκουσα χθε και στην Επιτροπή Αλία. Είπατε κάποιε φορέ ότι μιλάτε με, από προσωπική πλευρά περισσότερο παρά ω ε, πρόεδρο ε, του Συμβουλίου και αυτό ήταν μια ανακούφιση για μένα, για να είμαι μετά από πολλούς υπουργού που ήρθαν εδώ και ε, χρησιμοποίησαν τη γλώσσα του Συμβουλίου για να κρύψουν ε, την προσωπική τους άποψη. Για την κοινή αλληλευτική πολιτική ε, έχουμε ήδη ψηφίσει για σημαντικές, ε, σε άλλες επιτροπές έχουμε ψηφίσει, όμως στη δική μας είχαμε 50 ψήφους υπέρ κατά μηδέν για την σημαντική μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ε, κοιτάζω εδώ και προς τους συναδέλφους του ΑΕΛΚΑ ε, για να μας βοηθήσουν και στην ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα σε δύο εβδομάδες για να διασφαλίσουμε μια πραγματική ισχυρή ε, θέση διαπραγμάτευσης για το Κοινοβούλιο. Ίσως μπορείτε να σχολιάσετε αυτό λοιπόν. Νομίζετε ότι αν ε, υιοθετήσει το Κοινοβούλιο σε δύο εβδομάδε ε, την θέση της, ε, της, της Επιτροπής Αλληλευτικών Υποθέσεων. Αυτό θα διακινδυνεύσει ε, την, το μέγεθος και την έκταση της ε, μεταρρύθμισης αυτής. Επιπλέον, κάτι άλλο που βρίσκεται στο θεματολόγιο σας, ε, την ανάγκη να επιληθούν ε, τα ζητήματα που υπάρχουν για τα μακροπρόθεσμα ε, σχέδια διαχείρισης, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ στο μέλλον. Και δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόταση. Αν κάποιος δεν μπορεί να δείξει ποια είναι τα πρακτικά βήματα που μπορούν να γίνουν για να προωθηθεί το ζήτημα αυτό, τότε οι συντονιστέ είπαν ότι ίσω ε, πρέπει να εμποδίσουμε, να μπλοκάρουμε την μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Ξέρω ότι κανένα δεν το θέλει αυτό και ελπίζω ε, να μα δώσετε κάποια μικρά στοιχεία που θα μα βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ, Chris Davis. Έτσι κλείνουμε τον κύκλο των ε, συντονιστών. Ε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις ε, ερωτήσεις σας. Πρώτα της Bridget για το greening, αυτή την οικολογική διάσταση, το πρασίνισμα στην ε, κοινή γεωργική πολιτική. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ε, ισχυρή τέτοια οικολογική διάσταση στην μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής και αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βεβαίως μπορώ να σα δώσω την επίσημη θέση, δηλαδή το Συμβούλιο δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμα τη θέση του για το greening, όμως αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι κινούμεθα προ ένα συμβιβασμό αυτή τη στιγμή που θα βασίζεται στην πρόταση της επιτροπή, Δηλαδή, το πρασένισμα του πρώτου πυλώνα. Και να εργαστούμε με τα τρία κριτήρια που έχει καθορίσει ε, η Επιτροπή για να ε, θεωρείται επιλέξιμος ένας ε, γεωργός για ενισχύσεις του greening. Έχει συζητηθεί αυτό επί μακρόν. Πρέπει να δούμε αν θα εξετάσουμε άλλους πιο ευέλικτους τρόπους ε, για να καθίσταται κάποιος επιλέξιμος για το greening, γιατί ας πούμε η Κύπρος και η Σουηδία είναι πολύ διαφορετικές χώρες ό,τι αφορά τα γεωργικά του συστήματα, το μέγεθος των καλλιεργειών και ούτε καθεξής. Εξίσου διαφορετικές είναι και όλες οι χώρες ανάμεσά τους. Επομένως, όταν ε, προσπαθούμε να ορίσουμε μια κοινή πολιτική ε, σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ούτω καθεξής, πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξία από χώρα σε χώρα. Όμως, ταυτόχρονα, από πλευράς greening θέλουμε να υπάρχει μια ισοδυναμία, να υπάρχουν κοινά πρότυπα ε, στα όσα θέλουμε να εφαρμόζουν και να υλοποιούν οι γεωργοί ε, σε ό,τι αφορά την οικολογική διάσταση για να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Τέλο πάντων, αυτή η συζήτηση συνεχίζεται για πολύ καιρό τώρα. Υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει. Ε, υπάρχει πρόταση για μεγαλύτερο κατάλογο ε, για τι επιλογέ των χωρών ε, που συμπεριλαμβάνονται, για να μην υπάρχουν τρία πολύ αυστηρά κριτήρια. Η Επιτροπή αυτή έχει προτείνει ένα τέταρτο κριτήριο, αλλά θεωρώ ότι μάλλον θα εστιαστούμε στην πρόταση της Επιτροπής αυτή θα είναι η βάση μας για την τελική θέση του Συμβουλίου. Όμως θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις για τους τρεις διαφορετικούς ε, τομείς. Για ζητήματα όπως ε, ε, το ζήτημα της, ε, της ποικιλία ε, των των καλλιεργειών. Ξέρω ότι εσεί είχατε προτείνει την ε, αμυψησπορά. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ε, προτάσεις ε, για, για να τεθεί βάση μεμονωμένη καλλιέργεια και πρέπει να δούμε τι είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών σε κάθε χρόνο. Αλλιώ. θα πρέπει να γίνεται εκτίμηση ετησίω. Ε, με βάση την καλλιέργεια που υπάρχει στο αγροτεμάχιο και σε ποιο σημείο του κύκλου αμυψησποράς βρίσκεται αυτή η καλλιέργεια. Και αυτό είναι ε, τρομερά γραφειοκρατικό βεβαίως. Νομίζω λοιπόν ότι η διαφοροποίηση η εμψησπορά θα είναι κάτι προτιμότερο ε, σε σχέση με την διαφοροποίηση των καλλιεργιών σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο ε, στο, στο έδαφος. Όμως, ό,τι αφορά τη διαχείριση, η, διαφοροποίηση των καλλιεργιών είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί και να τύχει διαχείριση. Νομίζω ότι η, Επιτροπή, λοιπόν, η πρόταση τη Επιτροπή μπορεί να αλλάξει σε ό,τι αφορά την διαφοροποίηση. Ήδη έχει υπάρξει μια πρόταση, δηλαδή το κατόφλι πάνω από το οποίο απαιτούνται τρει καλλιέργειε σε ένα αγροτεμάχιο είναι τα τέσσερα εκτάρια. Πρέπει να αυξηθεί. Ξέρετε λοιπόν ότι το να, καλέ, το να ζητήσουμε από έναν αγρότη που έχει τέσσερα εκτάρια να έχει τρει διαφορετικέ καλλιέργειε, ε, κατά πόσο ε, είναι λογικό ή όχι, το βλέπετε. Επομένω, ίσω μπορεί να αλλάξει, να αυξηθεί αυτό το όριο. Υπάρχει μια άλλη πρόταση και από το Κοινοβούλιο, όπου θα αυξηθεί η διαφοροποίηση των καλλιεργιών, να έχουμε ένα κατόφλι κάτω από το οποίο δεν υπάρχει προϋπόθεση και υποχρέωση διαφοροποίηση. Μετά να έχουμε ένα κατόφλι ενδεχομένω όπου να, απαιτούνται τουλάχιστον δύο καλλιέργειε και πάνω από αυτό τρει. Και έτσι να υπάρχει πρακτικά δηλαδή για τους γεωργούς που έχουν μικρή έκταση να, ε, να, με διαφοροποίηση, αλλά σε λογικά πλαίσια. Αυτή είναι η συζήτηση λοιπόν ε, που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή για την διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Τώρα, για κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, ε, περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος. Ε, είναι κάτι το οποίο είχε παραχωρηθεί στο, στο παρελθόν, δηλαδή πληρώναμε του γεωργού για να μην κάνουν τίποτα. Οι περιοχέ οικολογικού ενδιαφέροντος ε, τώρα θα αποτελέσουν ένα κριτήριο επιλεξιμότητα για να λάβει κάποιο επιδότηση. Όμω θα πρέπει κάτι να κάνει ο γεωργό με αυτή την, ε, ε, με αυτή την καλλιέργεια, με αυτή την έκταση, να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα οικολογικό όφελο. Δεν χρειάζεται να είναι αρρώσιμη η γη αλλά να αποτελεί περιοχή σημαντικού οικολογικού ενδιαφέροντος και αξίας. Επομένως υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση εδώ πέρα και η πρόοδος είναι σημαντική γιατί δεν μπορούμε να εστιαστούμε στην αγρανάπαυση μόνο και να, να μειώνουμε έτσι την αρρώσιμη γη μας. Αν συμβεί αυτό στο μέλλον, τότε θα πρέπει να γίνει αυτό για λόγους ε, βιοποικιλότητας ε, και οικολογικής αξίας. Τώρα, το κατά πόσο θα συμφωνηθεί το 7%, ξέρω ότι προτιμάτε το 10%, αυτή ήταν η πρόταση που είχε γίνει. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια αλλαγή σε αυτόν τον αριθμό. Μάλλον βέβαια προς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλετε εσείς και ίσως μπορεί να υπάρξει αύξηση. Και πάλι νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει σημαντικές ε, προτάσεις εδώ, ενδιαφέρουσες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε δηλαδή από έναν αριθμό, να, να κινηθούμε, να το αυξήσουμε στο μέλλον, παρά να προσαρμοστούμε αυτή τη στιγμή ε, στους χώρους οικολογικού ενδιαφέροντος. Αλλά και πάλι από προσωπικής άποψης ε, σας μιλώ αυτή τη στιγμή για να σας ενημερώσω για τη συζήτηση. Ε, στο τέλη Μαρτίου ελπίζουμε να, έχουμε τελική οριστική θέση και εκεί θα είναι ξεκάθαρη η θέση του Συμβουλίου, την οποία και εγώ θα πρέπει να περασπιστώ ως ε, πρόεδρος ε, του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τους μόνιμους ε, βοσκοτόπους, που είναι το άλλο κριτήριο επιλεξιμότητας, είναι ε, ένα ζήτημα ίσονος σημασία για τις περισσότερες χώρες. Έχουν πολύ μικρό ποσοστό μόνιμων βοσκοτόπων στη χώρα τους. Υπάρχουν ήδη περιορισμοί στο ποσοστό των βοσκοτόπων αυτών ε, αυτή τη στιγμή είναι 10%. Για την Ιρλανδία, για παράδειγμα, που το 85% της αρρώσιμης γης είναι μόνιμοι βοσκότοποι, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό συμβαίνει και στη Γαλλία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε Κάποιε πρακτικέ ε, λύσει ε, για να δούμε πώ μπορούμε αφενό ε, να προστατεύσουμε την αξία των μονίμων βοσκοτόπων αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει μια διαχείριση καλλιεργειών που απαιτείται. Θα δούμε και άλλες σημαντικέ και πολύτιμε καλλιέργειε στις... και αυτό μα αφορά και σε ό,τι φορά τι καλλιέργειε πρωτεϊνών που μπορούν να αξιοποιηθούν για να φτάσουμε στο ποσοστό που θέλουμε. Για την απλούστευση υπάρχει μια πραγματική αιμονή στο Συμβούλιο ε, σε ό,τι αφορά την ανάγκη απλούστευσης. Δεν θέλουμε όμως να υπάρχει μια διαδικασία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που θα, μας, ε, ε, που θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να επιθεωρήσουν και να ελέγξουν τις προποθέσει και θα είναι και κάτι, μια, μια τρομερή γραφειοκρατία και για τους γεωργού. Η αρχική πρόταση λοιπόν την οποία στήριξαν και στήριξε και το ελεγκτικό συνέδριο που εξέφρασε προβληματισμό για τη γραφειοκρατία και το κόστος ε, υλοποίησης της νέας ε, κοινής γεωργικής πολιτικής. Η τελική θέση λοιπόν του Συμβουλίου θα προσπαθήσει να καταστήσει όσο το πιο απλό το σύστημα για τους γεωργούς τους ίδιους αλλά και για τις χώρες. αυτό θα είναι μια συνολική ε, θέση και προσέγγιση που θα έχουμε για όλα τα ζητήματα. Αυξάνεται όμως και η εστίαση για την απλούστευση για τους υπουργού, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που θα πρέπει να υλοποιήσουν τη μεταρρύθμιση και να βρούμε τον τρόπο να γίνει αυτό στι χώρε μας. Τώρα, όσον αφορά την ε, πρόταση της Λίντα και τις ε, ερωτήσεις της για την κοινή πολιτική, τα κύρια ζητήματα εδώ είναι οι απορρίψει. Πώς θα σταματήσει αυτή η απαράδεκτη ε, πρακτική όπου ουσιαστικά ζητάμε από τους ε, αλληλείς ε, να απορρίπτουν τεράστιες ποσότητες ηχθείων γιατί δεν μπορούν να τις εκφορτώσουν. Έχουμε έναν άτλαντα στην Ιρλανδία, δηλαδή έχουμε εκτιμήσει στο δικό μας στόλο το την έκταση του προβλήματος των απορρίψεων και είναι τεράστια αυτή η έκταση. Σε πολλές, φορέ έχουμε απόρριψη 40% των αλληλευμάτων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Το μεγάλο θετικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ε, ΚΑΠ που ελπίζουμε να γίνει κατά τη διάρκεια της ε, θητείας αυτής, της κοινοβουλευτικής θητείας, αλλά και της ε, δικής μας Προεδρίας, είναι να γίνει μία ε, μεταρρύθμιση που θα συμφέρει, θα είναι προς το συμφέρον και της ε, βιομηχανίας αλλά και ε, των πολιτών που προβληματίζονται και ανησυχούν για το μέλλον της αλίας στην Ευρώπη. Ε, λοιπόν, μας αφορά λοιπόν το ζήτημα των απορρίψεων της μέγιστης της βιώσιμης απόδοσης και άλλων ζητημάτων αλλά ουσιαστικά δεν θέλουμε να σχεδιάσουμε κανόνε και μετά όλο αυτό να μα αποτελέσει ένα τεράστιο πονοκέφαλο, γιατί δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Αν εξετάσετε λοιπόν μια χώρα όπω η δική μου, έχουμε μικρό σχετικά στόλο, ναυτικό, εμπορικό ναυτικό. Ε, οι ταλαιαυτικά σκάφη ε, πιάνουν περίπου 20% του, των αλλιευμάτων και έχουμε τεράστιους πορτογαλικούς, ισπανικούς, ε, ό,τι θέλετε στόλους ε, στα υδατά μας κάθε μέρα και πρέπει να το επιβλέπουμε όλο αυτό. Αν λοιπόν ε, εισάγουμε μια τέτοια πολιτική, νέα κοινιαλευτική πολιτική χωρίς να λάβουμε υπόψη τον κλάδο αυτό θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε με το ε, Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή από πλευρά Συμβουλίου για να βρούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά μια πραγματική λοιπόν μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά τι ε, απορρίψει και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και να πάμε να κινηθούμε προ ε, μια περιφερειακή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, ούτω ώστε οι χώρε να μπορούν να παίρνουν αποφάσει σε περιφερειακό επίπεδο στην περιφέρεια όπου αλλιεύουν, αντί να έχουμε αυτές τις τεράστιες μακρόχρονες διαδικασίες ε, με τα θεσμικά όργανα. Για την κοινή αλληλευτική πολιτική, λοιπόν, ελπίζουμε ότι θα έχουμε θέση του Συμβουλίου ε, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου για τον Γενικό Κανονισμό. Ε, για το Ταμείο Ελληνίας αυτό θα γίνει περίπου τον Απρίλιο. Πρέπει να ξέρουμε τι μορφή θα λάβει το πολιετές δημοσιονομικό πριν συμφωνήσουμε. Και πάλι έχουμε μια παράλληλη διαδρομή με το Κοινοβούλιο εδώ σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που θα δώσει και την εντολή στο Κοινοβούλιο να διαπραγματευτεί στους τριμερείς διαλόγους. Επομένως, θα συγχρονιστούμε ουσιαστικά και βεβαίως ε, οποιαδήποτε στιγμή είναι τόσο φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα μας που μπορεί να ξεφύγουμε. Αν γίνει, θα γίνει. Ε, και οι Λιθουανοί συνάδελφοι θα προσπαθήσουν να συνεχίσει το έργο μας και μετά από τη Λιθουανική η Ελληνική. Ε, όμως ε, σίγουρα θα είναι όλο και πιο δύσκολη η οριστικοποίηση ε, της μεταρρύθμισης γιατί μετά έχουμε και ευρωεκλογέ ε, και νέα επιτροπή μετά από αυτό. Θα είναι πραγματικά τραγωδία λοιπόν αν δεν καταφέρουμε ε, να ολοκληρώσουμε, να συμφωνήσουμε την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και αλληλευτικής πολιτικής πέρα, τα, πέρα των πρακτικών προβλημάτων που θα διαμορφωθούν από το 2014 και μετά. Τώρα, για την θέση του Chris Davis ε, για το διοργανικό πρόβλημα, υπάρχει πραγματικά πρόβλημα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της, της συνθήκης της Λισαβόνας, σε ό,τι αφορά τις εξουσίες λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά τα πολιτή διαχειριστικά ε, προγράμματα για την αλληλεία. Και έχω δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσω να να συμβάλλω ώστε να σημειωθεί πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Το πρώτο μα συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα ω ε, βασικό και μόνο θέμα ε, κατά τη διάρκεια του γεύματο είναι αυτό το διοργανικό ζήτημα. Και το έχω πει ξεκάθαρα και πολύ ομά ότι θα είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχουν ισχυρές θέσει ε, στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις εξουσίες που προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνα. Ε, εξίσου ισχυρές και έντονες είναι και αντιδράσει και από το Συμβούλιο. Πρέπει να συγκεράσουμε και τις ε, δύο απόψεις ε, ως πολιτικοί για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα γιατί αυτό θα βοηθήσει και γενικά ε, το ζήτημα της μεταρρύθμισης της ε, πολιτικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, αυτά τα μπιφτέκια δεινού στα οποία αναφερθήκατε, είναι πηγή σημαντικού προβληματισμού και σημείο ενδιαφέροντος για τα ΜΜΕ και στην Ιρλανδία και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δεν το γνωρίζετε, έχουμε μια αρχή ασφάλειας ε, τροφίμων στην Ιρλανδία που συνεργάζεται με το Υπουργείο μου σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα αυτά της ε, επιστημική ασφάλειας, επισήμανσης κτλ. Ουσιαστικά εκείνοι τι κάνουν, παίρνουν δείγματα διαφορετικών προϊόντων του λιανεμπορίου και αυτό συστηματικά και τώρα ε, κάνουν ε, τεστ DNA σε αυτά τα ε, δείγματα για να δουν ακριβώς, να διακριβώσουν τι περιλαμβάνουν. Ορισμένα λοιπόν από αυτά τα δείγματα, στα φθηνότερα βέβαια από τα προϊόντα, είδαμε ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό ε, κρέατος αλόγου στα μπιφτέκια βοδινού. Κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό Υπάρχει λοιπόν ε, μια διαδικασία διαρεύνησης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά απαιτείται περαιτέρω δειγματοληψία και των συστατικών και των ίδιων ε, των προϊόντων. Το εργοστάσιο έχει σταματήσει την παραγωγή αυτή τη στιγμή και τα περισσότερα βέβαια από αυτά τα προϊόντα είχαν ε, ε, εξαχθεί προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό υπήρξε και σχέδιο και στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο που είχε ένα παρόμοιο ε, πρόβλημα με DNA διαφορετικών ε, κρεάτων μέσα σε αυτά τα πιφτέκια. Επομένω, βλέπουμε εδώ πέρα ότι όταν έχουμε πολύ χαμηλά ε, ποσοστά τέτοιων ε, συστατικών, αυτό μπορεί να εξηγηθεί και με άλλους τυχαίους ε, ε, τρόπους. Για το πώς δηλαδή έχει μεταφερθεί το προϊόν, όταν γίνεται ο έλεγχος DNA, ε, μπορούμε να εντοπίσουμε ελάχιστα ίχνη που να δείχνουν ότι μπορεί να υπήρξε ένα ζήτημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή στο σφαγείο ή οτιδήποτε άλλο. Αν όμως υπάρχει ε, πιο σημαντικό ποσοστό από τέτοιου ίχνους που φτάνει το 15-20% ε, ε, DNA ύπου ή βοδινού ε, σε αυτό το κρέας, τότε υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και χρειάζεται μια καλύτερη απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν διενεργείται αυτή η εξέταση αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι οι Ιρλανδικέ αρχέ έχουν έρθει σε επαφή με τι Βρετανικέ αντίστοιχε αρχέ για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση για να καθησυχάσουμε και του καταναλωτέ επ' αυτού, όμως να τονίσω το εξή δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας τροφίμων, είναι ζήτημα ιχνηλασιμότητας και επισήμανσης ε, για να διασφαλίσουμε ε, να καθησυχάσουμε του καταναλωτέ. Γιατί οι περισσότεροι καταναλωτέ τρώνε έτσι κι αλλιώ ε, κρέα αλόγου. δεν είναι ουσιαστικό το πρόβλημα. Μην δημιουργήσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα όταν δεν υπάρχει. Ε, Απλώ οι καταναλωτέ πρέπει να γνωρίζουν και έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι τρώνε και τι καταναλώνουν. Πρέπει λοιπόν ε, να διασφαλίσουμε ότι θα διαμορφωθούν συστήματα ελέγχου επισήμανσης και χνελασιμότητα για να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι καταναλώνουν. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Και ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον ε, θα μάθουμε ακριβώ τι συνέβη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Chris Davis για τις παρατηρήσεις του σε ό,τι αφορά την ε, συνάντηση της Επιτροπής χθες ε, επιβεβαιώνω τις δεσμεύσεις που έκανα και χθε ε, για την πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί στα διοργανικά ζητήματα, αλλά ε, και ότι απευθύνω έκκληση και στη δική σα Επιτροπή και σε άλλους βουλευτέ να συνεργαστείτε με την Ιρλανδική Προεδρία για το ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων κοινή γεωργικής και αλευτικής πολιτικής μέχρι τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Φτάνουμε στον δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Η κυρία Άουκεν έχει ζητήσει το λόγο. Θα, μιλήσω, θα αναφέρω τα ονόματα. Η Dagmar Rockparent. Frau Schilders, Schnellhardt, Herr Gebrandi, Frau und Frau ξέχασα κάποιον. Παρακαλώ. Όχι, βρίσκεσαι στον κατάλογο. Ιδιαίτερα όσον αφορά την επισήμανση των προϊόντων, νομίζω ότι συχνά είμαστε πιο αυστηροί με τις ζωοτροφές παρά με τα δικά μας ε, τρόφιμα. Είναι μια συζήτηση την οποία νομίζω πρέπει να έχουμε και εδώ, αλλά και γενικά. Η κυρία Ροτμπέρεντ, ευχαριστώ πολύ Ματίας, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία ε, λόγια του Προέδρου μας ε, ήταν πολύ σωστά. Είμαστε πιο αυστηροί με την ε, επισήμανση. Μιλάω αγγλικά για να μην χρειάζεται τα ακουστικά σας, αλλά μπορώ να μιλήσω και γερμανικά αν θέλετε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας, Της γλώσσας. Είμαστε λοιπόν πολύ αυστηροί όσον αφορά τις ζωοτροφές μετά την σπογγόδια εγκεφαλοπάθεια των βοηδών. Ε, οι εμπειρίες μου τα τελευταία 23 χρόνια στο Κοινοβούλιο αλλά και στον τομέα της επισήμανσης και της προστασίας της υγείας του καταναλωτή και της υγείας των ζώων είναι ότι μόνο σε περίπτωση κρίσης ε, ξαφνικά τα κράτη-μέλη γίνονται απαλή, απαλά βελούδο. ε, σχεδόν ε, ε, ξεγλιστράνε μέσα από τα χέρια κανενός. Όσον αφορά λοιπόν ε, την επισήμανση, ε, δεν αναφέρεται κάθε συστατικό και δεν ήμασταν πολύ... δεν είχαμε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την επισήμανση, διότι από την άλλη μεριά του Κοινοβουλίου μου είπαν ότι ε, και τι θα γράφουμε πάνω στα σαλάμια. Ε, και τώρα μιλάμε για τα πιφτέκια. Και, ε, πρέπει να πω και πραγματικά πρέπει να πω ότι ε, υπήρξε τέτοια μείωση της κατανάλωσης των πιστακιών σε όλη την Ευρώπη που θα ε, υπάρξει αντίδραση. Εσείς ε, μιλάτε για την ασφάλεια του προϊόντος, λέτε ότι δεν επηρεάζεται η ασφάλεια. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η επιλογή του καταναλωτή. Και θα ε, διαπιστώσετε υπάρχουν μεγάλες ομάδες ε, θρησκευτικές ε, που αρνούνται να φάνε κρέας αλόγου λόγω της θρησκείας τους ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση να έχουμε περισσότερους που αρνούνται να φάνε χοιρινό. Ε, είτε επειδή δεν τους το επιτρέπει ε, το, ε, η θρησκεία τους ή επειδή δεν θέλουν να φάνε χοιρινό. Ελπίζω... λοιπόν, να γίνει κάτι όπως έγινε πριν 20 ε, χρόνια που βρεθήκανε σκουλικάκια στα ε, ψάρια και ξαφνικά είχαμε ε, νομοθεσία για την υγιεινή των ψαριών ότι πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία 5 ή 10 λεπτά μετά την αλία το ψάρι. Μπορεί να μην το θυμάστε, ήταν τεράστιο θέμα πάντως και όχι μόνο στη Γερμανία, παντού. Και βρήκαμε αυτά τα σκουλικάκια τα οποία δεν ήταν θέμα ασφαλείας του καταναλωτή αλλά είχε αδειάσει τόσο πολύ ο κόσμο που έπρεπε να κάνουμε κάτι. Και το ίδιο ακριβώ συνέβη με τη σπογγόδια ε, ε, εγκεφαλοπάθεια. Ξαφνικά είχαμε ένα ε, καλό σύστημα επισήμανση. Ελπίζω λοιπόν το θέμα των πιφτεκιών των βοδινών κάτι να γίνει όσον αφορά την πλευρά του καταναλωτή. Διότι εάν ε, δεν ε, κάνουμε κάτι για την επισήμανση, ανοίγουμε τις πόρτες ε, σε όλους να εξαπατήσουν τον καταναλωτή. Διότι, ναι, μπορεί να βάλει κανείς ό,τι θέλει κανείς σε εκεί βοδινό τρία χρόνια ήσασταν μέρος, μέλος του Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε λοιπόν πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Ίσως ε, λοιπόν ε, τώρα ως Προεδρεύων του Συμβουλίου ε, μπορεί να θέλετε να κάνετε, να κάνετε κάτι και να υποβάλλετε μια πρωτοβουλία για το πώς μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη επισήμανση. Ε, ερώτηση μιλούσατε σοβαρά, το εννοούσατε σοβαρά όταν ε, μιλήσατε για τις ε, διαφορές ε, στην κοινή γεωργική πολιτική. Είμαι ευγνώμων προς τη Λίντα που θύμισε σε όλους ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή δεν είναι ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Απέχει έτη φωτός. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο με πολύ μικρή διαφορά και οποιονδήποτε συμβιβασμό ψηφίσει ε, η Επιτροπή Γεωργίας μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι δεν θα είναι η ίδια ψηφοφορία με, του, με όσον αφορά τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και την αμυψησπορά. Εσείς αναφέρεστε στην ποιότητα του εδάφους, ε, να είμαι πιο συγκεκριμένη. Ναι, μας ενδιαφέρει η ποιότητα του εδάφους, ε, μας ενδιαφέρει η λιγότερη κατανάλωση ε, φυτοφαρμάκων. και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να αυξηθεί η κατανάλωση. Γνωρίζετε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Το παλιό καιρό κάθε γεωργό ε, θα ε, ε, εφήρμοζε την ανυψισπορά, διότι ήταν καλή γεωργική πρακτική. Εσείς όμως είπατε ότι είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί η άμεψη σπορά και θέλουμε να, πώς το είπατε, να την εφαρμόσουμε εύκολα και να έχουμε ένα απλό σύστημα, πιο φτηνό. Σωστό αυτό, αλλά εάν πούμε ότι με την ε, άμυψη σπορά μπορούμε με υπέρυθρες ακτίνες να δούμε αν υπάρχει ε, αμυψισπορά, ε, ε, εάν πιστεύουμε ότι το μισό των γεωργών ε, θέλουν να μας εξαπατήσουν, που ελπίζω να μην είναι η, η περίπτωση. Ε, αυτή πράγματι είναι η καλύτερη προσέγγιση και θα μπορούσα να συμφωνήσω όσον αφορά την διαφοροποίηση, αλλά θα πρέπει να επιμείνετε στο θέμα αυτό και όσον αφορά τη, τον αριθμό των καλλιεργιών στα, στις διάφορες εκτάσεις. Εάν ε, όμως ε, μιλάτε για κάτι τέτοιο σε τεράστιο αριθμό εκταρίων, ε, δεν συμφωνώ μαζί σας και φοβάμαι ότι και άλλοι δεν θα συμφωνήσουν. Επίσης, φοβάμαι ότι όσον αφορά την επιβολή του νόμου, μάλλον επιλέγουμε υπερβολικά εύκολες λύσεις. Εσείς είπατε ότι θέλετε να ξεκινήσετε τον τριμερή διάλογο πάνω στην ε, ηλεκτρονική ε, ε, ταυτοποίηση των βοηθών. Εμείς χάσαμε την ευκαιρία εδώ στο Κοινοβούλιο να έχουμε υποχρεωτική τέτοια ταυτοποίηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε υποχρεώσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ηλεκτρονικό σύστημα ανιχνευσιμότητας των βοηθών. Δεν το κάναμε αυτό. Ε, εάν λοιπόν πιστεύουμε ότι είναι πιο εύκολο να γίνει με διαφορετικό τρόπο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και μέσω τη κοινή γεωργική πολιτική. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε συνεπεί, θα πρέπει να ε, ελέγχουμε και να εφαρμόζουμε τα πράγματα απλά σε όλου του τομεί. Όσον αφορά λοιπόν ε, την μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, φοβάμαι ότι ε, αν πιστεύετε ότι τόσο μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού του 40% μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, με τρόπο απλοποιημένο, ε, να εφαρμοστεί με τρόπο απλοποιημένο, τότε να δώσουμε μια λευκή επιτυχία στα κρατη και να του πούμε κάντε ό,τι θέλετε, διότι αλλιώς θα αποτύχετε. Τουλάχιστον με τις ε, ε, προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιτάπητος. Επανέρχομαι σε μια τελευταία παρατήρηση και κατόπιν θα κλείσω, Ματία, σε ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ. Ε, Θέλω να αναφερθώ στα ψάρια και στις απορρίψεις. Συμφωνώ ότι έχουμε πρόβλημα εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα απορρίψεων σε κάθε αλίευμα. αλλά επιτρέπουμε έτσι λίγη περισσότερη ευελιξία ε, κατά την αλληλεία. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό εάν απλά αλλάξουμε το μέγεθος των δικτύων του ματιού δηλαδή. Ο Κρι Ντέιβις ε, δεν είναι πια εδώ. Σίγουρα θα συμφωνούσε αμέσως, ε, Καθώ και άλλοι θα συμφωνούσαν. Ε, έχουμε την παλιά συζήτηση σχετικά με το μέγεθος του ματιού των δικτύων. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφο που Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω σήμερα εδώ. Επίσης, ε, χαίρομαι που απαντήσατε με τόσες λεπτομέρειες ε, στις ερωτήσεις μας σε έξι μήνες. Ελπίζω και εγώ να τα καταφέρω εξίσου καλά με εσά κατά τη διάρκεια της δικής ε, της Προεδρίας Λουθανίας. Μιλήσατε για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το διοικητικό ε, τμήμα και άχθος σε ό,τι αφορά τους ε, γεωργούς. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, ήδη υπάρχει σημαντικό διοικητικό άχθος για τους γεωργούς. Από την άλλη, ίσως οι γεωργοί είναι σε καλύτερη θέση να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει με το έδαφος, με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή με τις δασικέ εκτάσει. Επομένω. ίσως εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε στο ECF, γιατί είναι αλήθεια ότι η κάθε χώρα έχει και το δικό της ορισμό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας ε, σε ό,τι αφορά αυτή τη νέα τάση που βλέπουμε ότι το διοικητικό άχθος συνεχώς και αυξάνεται για τους γεωργούς. Το άλλο μου ερώτημα αφορά και πάλι την κοινή, ελευτική πολιτική, γεωργική πολιτική και το greening, την οικολογική διάσταση πρασίνισμα. Το, έχουμε μιλήσει πολύ για αυτό το ζήτημα, έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά είναι πολύ πιθανό, εάν ε, οι γεωργοί δεν συμμορφωθούν ε, με τις προϋποθέσεις ε, του greening, να μην λάβουν ένα τμήμα του του επιδόματος. Ίσως να υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν κυρώσει. Ε, κάτι άλλο που προβληματίζει και ανησυχεί τα βαλτικά κράτη είναι διαφορέ μεταξύ των, ε, των επιπέδων των άμεσων ενισχύσεων. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και μια δικαιοσύνη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να χαιρετήσω τον Υπουργό από τη χώρα μου και θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα κατά τη διάρκεια της Θέλω να αναφερθώ κι εγώ πάλι στο σκάνδαλο του κρέατος αλόγου στα μοσχαρίσια μπιφτέκια. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το πρόβλημα. Προσπαθήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσουμε μια πολύ φιλόδοξη νομοθεσία περί επισήμανσης, ε, έναντι ε, και κόντρα στις πιέσεις ε, των πολύ ισχυρών λόμπι. Ήταν μια πολύ φιλόδοξη νομοθεσία που δεν κατάφερε να περάσει βεβαίως άθικτη αλλά με συμβασμούς. Ας το σκεφτούμε λοιπόν όλοι τι έγινε. Όπως είπε και ο υπουργό, μόλις το 99% του μπορεί να ανοιχνευθεί στη χώρα προέλευσης. Άρα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε ευρωπαϊκά, εν μέρει αποτύχαμε. Και να ρωτήσω κάτι για την αλία και το θαλάσσιο περιβάλλον. Σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία μικρών αλληλευτικών κοινοτήτων ποια είναι η αποψή σχετικά με, την, ε, με τους στόλους στις μικρές παράκτες περιοχές. Ευχαριστώ, Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ε, Υπουργέ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος ε, με τις σαφείς απαντήσεις σας. Ε, άλλωστε γνωρίζετε πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ στο Κοινοβούλιο όσον αφορά το πρασίνισμα, την περιβαλλοντική διάσταση. Ήδη υπόθηκαν πολλά, αλλά οι δικοί μου γεωργοί λένε ότι αν ε, έχουμε τόση γραφειοκρατία, τότε θα τα παρατήσουμε, διότι είναι ε, σημαντική η... Ε, διότι είναι σημαντικό το άχθος. Γι' αυτό επικροτώ τις προσπάθειές σας για περισσότερη ευελιξία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τον κατάλληλο δρόμο. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβάλλουμε υπερβολικά μεγάλο άχθος υπόθηκε και οι γεωργοί το ξέρουν. Όταν η Κομισιόν ε, λέει ε, το 70% ε, να είναι ένα προϊόν, τότε ήδη έχουμε διακόψει την άμυψη σπορά. Όσον αφορά τα μπιφτέκια. το, το, να είναι νοθευμένα είναι παρανομία. Δεν χρειάζεται να έχουμε πιο ε, αυστηρούς κανόνες. Ε, πρόκειται για απάτη και πρέπει να υπάρξει ε, δίωξη. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους βρίσκει το δρόμο της η για την ε, ε, υγεία των ζώων. Αν το έχουμε αυτό τέλη Μαρτίου, δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να βρούμε μια καλή προσέγγιση ώστε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Δύο πράγματα μας ενδιαφέρουν. Καταρχήν τα τέλη για τους επίσημους ελέγχους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό και επιτρέψτε μου να αναφέρω. Ίσως έχετε κι εσείς ε, κάποια ε, ιδέα. Υπάρχει ε, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα τέλη, κατά 100-200% ακόμα και σε περιοχές που απέχουν 50 χιλιόμετρα η μία από την άλλη. το θέμα λοιπόν είναι μήπως δεν έχουμε ρυθμίσει αρκετά ή μήπως έχουμε ρυθμίσει υπερβολικά τα πράγματα. Ε, κατά τις εργασίες ε, για τον κανονισμό αυτό υπήρχαν και δύο άλλες προτάσεις. Ε, τα τέλη να πληρώνονται μέσω των φόρων ή αναζώο να καθοριστεί ένα ποσό και να λέμε ότι η κάθε διοίκηση μπορεί να ε, το αυξήσει να το μειώσει κατά 20-30% επειδή ε, είναι διαφορετικό το επίπεδο των μισθών λοιπά στην κάθε χώρα. Αλλά ε, ίσως να μπορέσουμε να βρούμε μια καλύτερη λύση ε, και να αποφύγουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το δεύτερο θέμα είναι η επίσημη έλεγχη κρέατος. Έχουμε διαπιστώσει ότι η παρούσα μορφή των ελέγχων ε, δεν ε, μας επιτρέπει τον εντοπισμό ζωονόσων και δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε λίγα λόγια σχετικά με το τι προτείνει η Επιτροπή ή το τι σχεδιάζει το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και σημαντικό για μένα είναι κατά τη συζήτηση αυτών των θεμάτων να επιδιώκουμε περισσότερο δημόσια συζήτηση. Ε, ίσως και από πλευρά του Συμβουλίου καλό θα είναι να ε, οργανωθεί κάτι τέτοιο ώστε να ξεκινήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Αναφερθήκατε και στην ε, μη ε, εμπορική εκτροφή ζώων. Ε, Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά καλά. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά θα ήθελα να πω και στους συναδέρφους μου εδώ που ε, συμμετείχαν στη συζήτηση. Ε, με αυτά που προβλέπονται όσον αφορά τις κατεξοδότηση πράξης, δεν μπορούμε ε, να μετακινηθούμε, διότι το Κοινοβούλιο θέλει να έχει λέγει και αφότου ε, ολοκληρωθεί το νομοθέτημα αυτό. Εσείς ε, ως Συμβούλιο βέβαια μπορείτε να καταψηφίσετε μόνο αν έχετε ομοφωνία, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να μετακινηθεί το, το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό, διότι όλες οι, απόψεις, ε, όλες οι ε, πλευρές είναι της απόψης ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σνέλχαρτ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό για τη σημερινή του παρουσία στην Επιτροπή μας. Όταν να μπήκε σε ισχύ η συνθήκη Λισαβόνας είχα την αίσθηση ότι επιτέλους και η αλληλευτική και η αγροτική πολιτική τα συμφέροντα, δηλαδή θα, λάβουν υπόψη τα συμφέροντα των 500 εκατομμυρίων πολιτών και όχι μόνο των άμεσα ενδιαφερομένων. Των αλλιέων και των αγροτών εννοώ. Ειλικρινά ε, μπορώ να πω με περηφάνεια ότι αυτό που κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την γεωργική και την αλληλευτική πολιτική, έχουμε κάνει πολλά πράγματα σε ό,τι μας ζητά η συνθήκη της Λαβώνας. Βεβαίως η Επιτροπή Γεωργίας κινείται κάποιες φορές σε στραβή κατεύθυνση και μάλλον να ενισχύει τα λόμπι του γεωργικού τομέα που έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των άλλων 490 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης. Ρωτώ. Ήδη έχετε ξεκινήσει ανεπίσημες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους βασικούς παίκτες της Επιτροπής Γεωργίας του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο για να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Επισήμως γνωρίζω ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Και δεν θα υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ανεπίσημα όμως τι γίνεται. Οι βασικοί παίκτες κλειδιά του Κοινοβουλίου και οι βασικοί παίκτες του Συμβουλίου μήπως ανεπισήμως έχουν αποφασίσει πώς θα δαπανηθούν αυτά τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη επταετία. Είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στην ε, Κύπρο και τη Σουηδία γεωγραφικά. Δίκιο έχετε, ναι. Άρα χρειάζεται και κάποια ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διαφορές. Οι χώρες όμω αυτές, όπως και όλες οι υπόλοιπες της Ένωσης, δυστυχώς ε, έχουν κάποιο κοινό στοιχείο. Φαίνεται να μην ενδιαφέρονται για τα κριτήρια που συνδέονται ε, με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά μόνο για την χρηματοδότηση. Δηλαδή, σαν ένα κουμπαρά, έτσι, ένα γουρνάκι κουμπαρά σε Βρυξέλλε, ε, που δίνει μόνο χρήμα και όχι ένα οργανισμό με συγκεκριμένου πολιτικού στόχου. Αν διαβάσετε για παράδειγμα τις εκθέσει ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, πραγματικά οδυνηρά είναι τα συμπεράσματα κανενό. Δηλαδή, Ελάχιστη τελικά είναι οι στόχοι που τελικά επιτυγχάνουν χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα κράτη-μέλη. Δείτε τα προγράμματα για τη γεωργία και το περιβάλλον. Είναι τόσο ευέλικτα που τελικά τα κράτη-μέλη μπορούν να τα εφαρμόσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ρέει το χρήμα στους αγρότες, χωρίς όμως κανένα όφελος ούτε για τη φύση, ούτε για το περιβάλλον εγώ δεν νομίζω τελικά ότι έτσι επιτυγχάνουμε του γενικότερου στόχου τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα προκειμένου. Κατανοώ ότι και οι αγρότε χρειάζονται μια κάποια ευελιξία. Δεν μπορούμε να του επιβάλλουμε μέτρα για το πρασίνισμα όπω αυτά προτείνει η Κομισιόν. Αλλά υπάρχει όμω και κάποιο άλλο λόγο για τον οποίο τα κράτη-μέλη επιζητούν αυτή την ευελιξία γιατί πολύ απλά δεν τους νοιάζουν τα κριτήρια, ούτε τα μέτρα για το πρασίνισμα, μόνο τα χρήματα θέλουν. Άρα πού, πού είναι η ισορροπία ανάμεσα σε μια α, ευελιξία που πρέπει να υπάρχει στα μέτρα μεν, αλλά όχι υπερβολική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν αυτή την ευκαιρία για τελικά να μην επιτυχάνουν κανένα στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής, απλά να γίνονται αποδέκτες χρημάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που συναντώ εδώ σήμερα ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καθώς και στους διερμηνείς και στους υπόλοιπους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου ευτυχία το 2013 και ένα εξαιρετικό πρώτο εξάμεινο το 2013 προς τον κύριο Υπουργό πιο συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά το κρέας ε, αλόγου έχουν υποθεί τα πάντα. Είμαι συγγήτρια για τον κανονισμό για την επισήμανση ε, του βόλιου κρέας. Κρέατος ε, πολλά έχουν υποθεί, δεν θέλω να πω κάτι. Το μόνο που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτό το ζήτημα που ε, προέκυψε στο, στην Ιρλανδία και στο Μένο Βασίλειο θέτει τρία ε, ζητήματα. Είπατε ότι δεν πρόκειται για ζήτημα δημόσιας υγείας, αυτό είναι σαφές. Όμως θεωρώ εξκανδαλώδες ε, να καταναλώνω ε, αλογίσιο κρέας, κρέας αλόγου όταν θεωρώ ότι τρώω βόδιο. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το ζήτημα για τους πολίτες μας. Και αυτό επιβεβαιώνει και την ε, σημασία φιλόδοξου ε, κειμένου για την επιστήμανση. Γιατί θα πρέπει να προστατεύει τους καταναλωτές και τους πολίτες, όμως θα πρέπει να σκεφτόμαστε και την ε, βιομηχανία, τον κλάδο δηλαδή, όσους κάνουν τη δουλειά τους σωστά, παράγουν προϊόντα του τομέα και του κλάδου σύμφωνα με τον νόμο αλλά παράλληλα υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που δεν του επιτρέπουν να καινοτομήσουν και να επενδύσουν. Πρέπει λοιπόν η νομοθεσία να είναι υπέρ και του καταναλωτή, αλλά και καλή την πίστη για του ε, εκπροσώπου ε, του κλάδου, για να του ε, προστατεύσουμε με την απαραίτητη νομική ασφάλεια. Δεύτερο σημείο για αυτό το πρόβλημα με το κρέας στην Ιρλανδία και το Βασίλειο υπάρχει και το ζήτημα του ελέγχου. Ξέρουμε όλοι ότι στα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες υπάρχουν προϊόντα που από πλευράς ποιότητας καθόλου δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια των κανονισμών μας και της νομοθεσία μας ή των απαιτήσεων των καταναλωτών. Έχουμε λοιπόν ένα, μια επαρκή απάντηση για αυτά τα προβλήματα. Και τέλος, ξέρετε το ζήτημα των τροποποιημένων οργανισμών, των γενετικώ μεταλλαγμένων οργανισμών. Ξέρετε λοιπόν ε, το ζήτημα και τη συζήτηση. Χθε εκπρόσωπος ε, ε, του Επιτρόπου Υγεία, ο Φρεντερίκ Βανσάν, είπε ότι στο άμεσο μέλλον η Επιτροπή δεν πρόκειται να υποβάλει αιτήματα ε, καλλιεργειών στα κράτη-μέλη. Βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβασμό μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Κρατών Μελών για τους, ε, για τους στόχους ε, της οδηγίας προβάλλοντας το ζήτημα των γενετικών τροποποιημένων οργανισμών. Ποια θα είναι όμως η θέση της Ιρλανδικής Προεδρίας σε ένα από τα ζητήματα που για μένα τουλάχιστον είναι εξαιρετικά σημαντικό και πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας ε, παράλληλα και την συνένεση μεταξύ κρατών μελών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και πρόεδρε Ματιάς. Ε, τι συμβαίνει με την κροατική καμπίνα. Ήθελα να ακούσω κροατικά. Αν μπορείτε δώστε μου τον αριθμό, γιατί ήθελα να τους ακούσω. Α, το 13. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η, κυρία Άουκεν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα μιλήσω πολύ σύντομα στα φτωχά αγγλικά μου. Να αναφερθώ στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Είμαι μέλος ε, της Επιτροπής Αναφορών ε, και την Δευτέρα ε, είχαμε το θέμα των μελισσοκόμων, διότι είναι αναγκασμένοι κατά κάποιους τρόπους ε, να χρησιμοποιούν ε, καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένες, ε, όχι για να αποφύγουν ε, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά για να αποφύγουν τα προβλήματα. Για τους μελισσοκόμους και για τους καταναλωτές και για τις μέλισσες δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλός ο τρόπος αυτός. Επειδή πολύ απλά δεν έχει κανείς τη βούληση να αποφύγει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στο μέλι. Στη γύρη δηλαδή. Σας ρωτώ λοιπόν, δεν θα μπορούσατε στην ε, όλη συζήτηση με τα βοηθή να λάβετε υπόψη σας και τις μέλισσες και τους καταναλωτές και τους μελισσοκόμους, ώστε να είμαστε βέβαιοι όταν αγοράζουμε μέλη όπου δεν υπάρχει επισήμανση ότι συμπεριλαμβάνει ε, γενικά τροποποιημένους οργανισμούς. να γνωρίζει ε, ότι δεν έχει τέτοιες ουσίες μέσα ο καταναλωτής. Ε, παρακαλούμε λοιπόν ε, το Συμβούλιο να φρενάρει την Επιτροπή που θέλει να δει το θέμα πολύ πρακτικά και να χειριστεί πολύ ελαφρά το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους. Κύριε Υπουργέ μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Well, uh, there was a lot of questions. Πολλές ε, οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όσο γίνεται, πιο εξαντλητικά. Για τα πρώτα ερωτήματα και τα σχετικά σχόλια για την επισήμανση θεμητά σχόλια. Πράγματι, ο καταναλωτή έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι τρώει. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή τροφίμων δεν έχουν κάποια απέτηση, δεν υποχρεούνται μάλλον να φέρνουν κάποια επισήμανση για τα επεξεργασμένα προϊόντα, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθεια για τη χώρα προέλευσης για κρέατα πέρα από το βόλιο κρέας ώστε και άλλες κατηγορίες ε, να μπουν στην ε, υποχρέωση για επισήμανση για τη χώρα προέλευση. Είτε είναι χείριο, είτε είναι πουλερικά, είτε είναι πρόβιο κρέας. Αλλά κοιτάξτε, εγώ μιλώ ως Ιρλανδός υπουργό Γεωργίας. Προτεραιότητα μας είναι να πάμε σε βάθος αυτής της υπόθεσης να δούμε πώς συνέβη αυτό το γεγονός πιστεύω ότι έχουμε πολύ αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης στην Ελλαδία. Οπότε και μόνο που έγινε αυτό το γεγονός και οι γενομικές μας αρχές χρησιμοποιούν ε, έλεγχο DNA δείχνουν πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό για μας και γενικότερη ποιότητα τροφίμων. Ο τομέας του κρέατος στην Ελλαδία ε, είναι πολύ ψηλά, γιατί είμαστε όχι μόνο η πρώτη η χώρα στον κόσμο που αναρωτιέται για τη χώρα προέλευσης, αλλά μετρούμε και το χνάρι ε, άνθρακα που αφήνει η κατανάλωση κρέατος φέρνος μόνο. 32.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις βόλιο κρέατος στην Ιρλανδία θα περάσουν από έλεγχο για τις εκπομπές ρήπων άνθρακα από την κατανάλωση βόλιο κρέατος πιο λοιπόν το χνάρι στον άνθρακα που αφήνει ε, το ίδιο το ζώο το οποίο εκτρέφεται με σκοπό τη χρήση του βόλου κρέατος. Κατανοείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για μας. Βεβαίως πάντοτε συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Ε, θεωρώ ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και το γεγονός ότι εξακριβώθηκε αυτή η υπόθεση λόγω των δοκιμών που κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Μας επιτρέπουν και να το συζητάμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Είτε λοιπόν ως υπουργό της χώρας μου, είτε ως ασκών καθήκοντα στο Συμβούλιο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για θέματα επισήμανσης για να αποτρέψουμε τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Τώρα, αν κατάλαβα καλά κάτι που είπατε πολύ συμφωνώ. Η θέση της Επιτροπής Γεωργίας δεν, του Κοινοβουλίου δεν αναγκαστικά θα είναι η ίδια με τη δική σας στην Ολομέλεια. Αλλά από και πέρα, εγώ το μόνο που να πω είναι ότι αυτό είναι δική σας υπόθεση, θα αποφασίσετε. Όταν δηλαδή το Κοινοβούλιο καταλήξει στην τελική του διαπραγματευτική του θέση για την ΚΑΠ, και το Συμβούλιο καταλήξει στη δική του δημοτική θέση, η δική μου δουλειά είναι να ηγηθώ των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα. Από εκεί πέρα εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στα θέματα τη Επιτροπή Γεωργία. Ήταν εσφαλμένο από πλευρά μου να σχολιάσω τις θέσεις επιτροπή Γεωργίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την διαφορετικότητα των καλλιεργιών έναντι τη αμφισπορά, η Κομισιόν επέλεξε την οδό τη διαφοροποίηση θεωρώντα ότι είναι μια μέθοδος που είναι πιο εύκολο και να υλοποιηθεί και να παρακολουθηθεί. Αυτό, από ό,τι γνωρίζω, είναι αποτέλεσμα εντονότατων συζητήσεων στην Κομισιόν υπέρ της μίας και της άλλης λύσης. Κατανοώ τα επιχειρήματα όμω και των δύο πλευρών. Και εγώ με το παρελθόν του αγρότη κατανοώ τα επιχειρήματα και των ΜΕ και των ΔΕ. Για το 40% του υπολογισμού, αυτό που υπόθηκε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι Ακόμα, με βάση τι προτάσει Κομισιόν και χωρί να έχουμε δει την τελική μορφή του πολιτού δημοσιονομικού πλασίου. τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βαθμιαία μείωση του ποσοστού του συνολικού προπολογισμού τη Ένωση για τη γεωργία. Με βάση την πρόταση επιτροπή ξεκινά από 38%. Όμω, η ΚΑΠ είναι το μόνο στοιχείο του πολιτισμού δημοσιονομικού πλασίου που δεν θα ε, συνυπολογίστε με βάση κάποιον δίκτυ. Ούτε δίκτυ πληροφοριοσμού, ούτε κανένα δίκτυ. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο για, την, ε, για το πολιετές οικονομικό πλαίσιο. Για όλους τους λόγους που και εσείς ε, αναφέρατε, αλλά και για λόγους ασφάλειας τροφίμων, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση έχουμε πραγματικά μια μεγάλη υποχρέωση να εγγυηθούμε ένα βιώσιμο και καινοτόμο σύστημα παραγωγής τροφίμων και μια πολιτική συλλογή δεδομένων στον Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το θέλουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε και τα χρήματα να το πληρώσουμε. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Σε ό,τι αφορά τις απορρίψεις, δυστυχώς, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το θέμα. Δεν αρκεί να αυξήσει το μέγεθο του ματιού του δικτυού. Ε, εν μέρει είναι μια λύση. Αλλά θα πρέπει να εγγυηθούμε ότι λαμβάνονται υπόψη και οι επιστημονικές θέσεις από την ε, ενδιαφερόμενη κοινότητα, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε τους γόνους. Πράγματι, οι γόνοι δεν θα πρέπει και γενικότερα τα ψάρια κάτω από ένα μεγέθο δεν θα πρέπει να αλλιεύονται και να μην μπαίνουν στην ε, ε, εμπορία. Το βλέπουμε ας πούμε, ακόμα και στις κελτικές ε, θάλασσες. Ε, εμείς το τελευταίο 12 είχαμε μία μείωση των απορρίψεων κατά 40% ακριβώ γιατί μεγαλώσαμε το μέγεθο του μαθητού του δικτύου. Είναι λοιπόν κομμάτι τη όλη στρατηγική. Αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα στην μεικτή αλεία. Δηλαδή το να αλλιεύει 3, 4 έως και 5 και 6 είδη α, ενήλικων στο ίδιο δίχτυ και το πρόβλημα τελικά είναι τι γίνεται με αυτό το μείγμα. Διότι μπορεί να έχουν το ίδιο μέγεθος και να τα αλλιεύει στο ίδιο βάθος υδάτων. Αλλά υπάρχει διαφορά από είδος σε είδος ε, και χρειάζεται λοιπόν να έχουμε τεχνικά μέτρα που να μας επιτρέψουν να επιλύσουμε εν μέρη πιστεύω αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να επιληθεί πλήρως. Θα υπάρχει το πρόβλημα λοιπόν του αλία που αλλιεύει ψάρια που δεν επιτρέπεται να τα αλλιεύει και αυτό είναι ένα απόφευκτο για το άμεσο μέλλον. Λέμε, αυξάνοντας ε, το μάτι του δικτυού και με άλλα τεχνικά μέτρα που αφορούν τα δίκτυα, εν μέρη βελτιώνουμε την κατάσταση, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα που δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να πούμε ότι μπορούμε να εξελίψουμε πλήρως τις απόρριψεις. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τη Λισαβόνα, με συγχωρείτε, θέλω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Πάντω χαίρομαι γιατί έχουμε πρόσωπο από τη Λιθουανία διότι η Ιρλανδία. Βεβαίω, ε, σε ό,τι αφορά την Προεδρία του Συμβουλίου, είναι μέρο μια τρόικα, λέει ο μιλητή. Είμαστε μέρο μια ομάδα τριών Προεδριών, Ιρλανδία, Λιθουανία και Ελλάδα, που από κοινού έχουμε ορίσει ένα πρόγραμμα. Οπότε θέλουμε να περάσουμε τη σκητάλη για κάποια ζητήματα που δεν θα καταφέρουμε να κλείσουμε στη Λιθουανία, όσο γίνεται όμω να περάσουμε πιο αμαλά και πιο εύκολα τα θέματα στη Λιθουανία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συνεργασία στο Συμβούλιο ανάμεσα σε αυτέ τι τρει χώρε. Κατανοώ αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο να κάνουμε κάτι πρακτικό και ρεαλιστικό για την ΚΑΠ, αλλά αυτή η ΚΑΠ και η μεταρρύθμιση τη να μην στοιχήσει υπερβολικά χρόνο και χρήμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του αγρότε. Πραγματικά προσπαθούμε και εμεί να επιφέρουμε την ισορροπία. Για τη δασοκομεία είπα τα σχόλιά μου και προσβλέπω στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν προκειμένου. Θέλουμε να δούμε ποια θα είναι η νέα κοινή προσέγγιση για τη δασοκομεία και την βιωσιμότητα αυτή. Αλλά και πάλι θα πρέπει να είναι κάτι ευνόητο και εύληπτο, ώστε να κατανοεί ο κάθε πολίτη τι του ζητείται να κάνει και σε ό,τι αφορά τι ιδιωτικέ εκτάσει, αλλά και τα δημόσια δάση, σε ό,τι αφορά το θέμα των βαλτικών χωρών ώστε να έχουν ένα ισότιμο μερίδιο στις άμεσες ενισχύσεις. Εγώ επισκέφτηκα και τις τρεις βαλτικές χώρες πριν από κάποιους μήνες για να έρθω σε επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς για τα ζητήματα αυτά. Τα εν λόγω κρατημέλη έχουν προσωπικά τη δική μου υποστήριξη και πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει και κάποια πρόοδο συζητήσεις για τα θέματα του πολιτισμοσονομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις ώστε η σε ένα εκτάριο. Στι βαλτικέ χώρε να έρθουν πιο κοντά στο μέσο όρο. Πιστεύω ότι έχει υπάρξει πρόοδο σε συζητήσει και με του υπουργού σα, αλλά και με τη δική σα βοήθεια εδώ στο Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα σχόλιά σα ε, για την ε, επισήμανση πράγματι το Κοινοβούλιο ήταν πάντα πολύ φιλόδοξο ό,τι αφορά αυτή την νομοθεσία και το Συμβούλιο θα συνεχίσει να εξετάσει τι εναλλακτικέ, λαμβάνοντα υπόψη για τι προτάσει τη επιτροπή των Έλθων. Αλλά δεν θέλω να υποσχεθώ πολλά εν Θέλω πρώτα και εγώ να δω ποιε είναι οι δυνατότητες στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι όμως το μέλλον ε, θα συζητήσουμε στο άμεσο μέλλον πάλι αυτό το θέμα, σε ό,τι αφορά πάλι την βιώσιμη αλληλεία και τη μεταρρύθμιση ελευτική πολιτικής. Μα αυτή είναι η, το όλο νόημα της μεταρρύθμισης. Θέλουμε βιώσιμε αλληλευτικέ κοινότητε, ταυτόχρονα με βιώσιμα αλληλευτικά αποθέματα ο καλύτερος τρόπος για να εγγυηθούμε βιώσιμη αλληλευτική κοινότητα σε 5-10 χρόνια ε, είναι να εγγυηθούμε ψάρια και στη θάλασσα. Ε, γι' αυτό δουλεύουμε τόσο πολύ σε θέματα μέγιστης ε, δυνατής απόδοσης και ανατεχνικά μέτρα. Σε ό,τι το πρασίνισμα. Ναι, χρειάζονται κάποιε νέε γραφειοκρατικέ απαιτήσει, αλλά θα το κρατήσουμε αυτό στο ελάχιστο. Το ελεκτικό συνέδριο μα ε, υπενθύμησε ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε τι δαπάνε χαμηλά. Σε ό,τι αφορά του επίσημου ελέγχου, περιμένουμε τι προτάσει τη Κομισιόν που θα έρθουν κατά πάσα πιθανότητα το Μάρτι, ώστε να καταλήξουμε σε μία θέση στο Συμβούλιο που ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε αυτές τις θέσεις του Συμβουλίου άμεσα μετά. Βεβαίως αυτό ε, σχετίζεται και με τις πράξεις αξιοδότηση. Σε ό,τι αφορά τα πολύ άμεσα σχόλια που ακούστηκαν για ποιες, τις, ποιες είναι οι ελπίδες του Κοινοβουλίου μετά την Λισαβόνα. Δέχομαι τα πιο πολλά από αυτά που είπατε. Δεν συμφωνώ με όλα πάντως. Δεν πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη και όλοι οι υπουργοί βλέπουν ε, τις Βρυξέλλες σε μια, αν θέλετε, μια αγροτικό κουμπαρά α, Δείτε πώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα σε σχέση με 20 χρόνια πριν. Έχουμε δραματικές αλλαγές. Η χνηλασιμότητα, για παράδειγμα, οι συνέπειε στην εφαρμογή διαφόρων οδηγιών, θέματα πολλαπλής συμμόρφωσης, ελέγχου, βιωσιμότητας. Και όλα αυτά έγιναν λόγω των μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ και λόγω των χρημάτων που επενδύουμε στην ΚΑΠ ώστε πραγματικά αυτά τα χρήματα να έχουν ένα νόημα. Πιστεύω ότι αυτή τώρα η μεταρρύθμιση θέλει να φέρει εξυγχρονισμό στην ό, στον όλο αυτό τρόπο σκέψη, ώστε να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει που δεν συζητήθηκαν ενεργά στην τελευταία μεταρρύθμιση όπω είναι ασφάλεια τροφίμων, ε, η βιοπικιλότητα, η βιωσιμότητα, αλλαγή του κλίματο. και γι' αυτό βλέπετε τις αλλαγές, τις προτάσεις στο δεύτερο πυλώνα της ε, ΚΑΠ, στην ε, ανάπτυξη τη της, ε, ανάπτυξη. Και βεβαίω και εγώ να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ε, βιάζεστε να μάθετε κροάτικα. Αυτό δείχνει και το μέλλον. Βεβαίω, βλέπω ότι ταυτόχρονα ότι πολλοί κάνουν καταβάλουν προσπάθεια να μιλήσουν αγγλικά και εγώ. Και εγώ μιλώ αγγλικό, αγγλικά και μόνο, αλλά θα πρέπει να καταβάλω την προσπάθεια να μάθω και άλλε γλώσσε. Για του γενικά τροποποιημένου, ξέρω ότι έχετε συγκεκριμένη θέση προκειμένου και δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο στο τομέα αυτό ε, στο Συμβούλιο, διότι δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ειδική πλειοψηφία. Αυτό που μπορεί να κάνει η Προεδρία είναι να αξιολογήσει κατά πόσον η στάση αλλάζει ή έχει αλλάξει. Ποιε είναι οι θέσει λοιπόν των κρατών μελών, να δούμε αν έχει αλλάξει ο συσχετισμό δυνάμεων, αλλά από και πέρα να και στην Κομισιόν να υποβάλει νέε προτάσει ε, με νέο σκεπτικό, ώστε να αλλάξει, ε, αν θέλετε, και η ψήφο των κρατών μελών. Αν τελικά θέλουμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο γιατί μιλάμε για γενετικά τροποποιημένο, θα πρέπει από τη μία να διασφαλίσουμε την ακυριότητα της ιστορικής αγοράς και να τηρούμε την αρχή της επικουρικότητας. Τέλος, για τις μέλισσε. Ο πληθυσμό των μελισσών αντιμετωπίζει κάποια πίεση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και αυτό αφορά κάποιες ασθένειες αλλά και οφείλεται και στην ανησυχία από τη χρήση κάποιων εντομοκτώνων. Και ανησυχίες όσο υπάρχουν λόγω των γενικά τροποποιημένων. Μπορούμε να πούμε ότι και αυτό είναι κομμάτι της συναπόφασης, δηλαδή η Επιτροπή σας θα πρέπει να προβεί στην δική της γνωμοδότηση ακριβώς για το θέμα που θέσατε. Άρα, ο πρώτος στον οποίο μπορείτε να αποτανθείτε για αυτές τις ανησυχίες σας είναι η επιτροπή σας. Να καταλέξετε σε μια θέση που να σας ικανοποιεί, ώστε μετά να αρχίσετε τις συζητήσεις με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν, για να μπορέσει να καταλήξει κάπου αυτή η πρόταση. Αυτά. Ήταν πολλά και ποικίλα αυτά που ακούστηκαν. Δεν ξέρω αν κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Όσο προσοχή, ξέρω ότι μας πιέζει και ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάντως για το ενδιαφέρον σας και αν θέλετε να απευθυνθείτε άμεσα σε μένα ως ασκούντα τα καθήκοντα του Πρόεδρου του Συμβουλίου ή σε μένα προσωπικά, με χαρά να ακούσω τι τις θέσεις και προσβλέπω στη μετέρα συνεργασία μαζί στο επόμενο εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την δυνατότητα της ανταλλαγής απόψεων μαζί σας. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλός ο διάλογος που μόλις είχαμε. Βλέπουμε όμως ότι είναι και πολύ ενδιαφέροντες καιροί, διότι μας περιμένει η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Ε, πολλή δουλειά μας περιμένει. Θα πρέπει να είμαστε και συνεννόηση μεταξύ μας. Ε, πρόκειται για δύο τομείς ε, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε λοιπόν τώρα την βασική δοκιμή μετά τη Λισαβόνα. Τελικά θα πρέπει να μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό τον οποίο να μπορούμε να δεχτούμε όλοι. Και γι' αυτό έχετε και εσείς, έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη ευθύνη. Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη. Νομίζω θα σας χρειαστεί και σας ευχαριστώ θερμά που απαντήσατε στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Και βέβαια αυτό που είπατε εσείς ισχύει και για σας, ε, ότι αν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε μπορείτε να πάσα στιγμή να έρθετε σε επαφή με τους συναδέρφους. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στη συνεργασία. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον επόμενο ε, υπουργό που βρίσκεται μεταξύ μας, ε, τον Υπουργό Υγείας της Λιθουανίας, της επόμενης δηλαδή Προεδρίας. Ε, σας καλωσορίζω θερμά. Και τώρα έχουμε να συζητήσουμε την έκθεση ε, του συναδέλφου Ούλμερ. Προτείνω λοιπόν ε, μία σύντομη εισαγωγή στην έκθεση, διότι αλλιώ θα έχουμε πρόβλημα χρόνου. Κύριε Ούλμερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι σχετικά σύντομο. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τεχνική έκθεση. Κυρίω ε, το θέμα είναι να ε, ε, μαζέψουμε σε ένα νέο κανονισμό τους ε, κανόνες που ισχύουν μέχρι τώρα και τους όρους της συνθήκης Euratom. Είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε μόνο κάποια, κάποια από τα άρθρα. Στην αιτιολογική έκθεση έχω γράψει τα περισσότερα που ήθελα να πω. Έχουμε επικαιροποιήσει λοιπόν ε, τις ε, ρυθμίσεις όσον αφορά τις ιονίζουσες ακτινοβολίες ε, και την προστασία των ανθρώπων από την ακτινοβολία αυτή. το θέμα είναι να αποφύγουμε την ακτινοβολία, προστασία σε περίπτωση που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε τελείως. γνωρίζω πολύ καλά τον τομέα αυτόν, διότι ε, επί 30 χρόνια στην ε, Γερμανία έχω εργαστεί ως ε, γιατρός ειδικά στον τομέα της προστασίας από την ακτινοβολία. Έχουμε πολλές νομικές πράξεις της Euratom και στην παρούσα πρόταση εφαρμόζουμε πολύ καλά τους στόχους της Euratom. Και έχω προτείνει σημαντική τροποποίηση στην ε, έκθεση. Ε, θα ήθελα να διαγραφεί τελείως το κεφάλαιο 9. Θα ήθελα το κεφάλαιο αυτό να συμπεριληφθεί σε ξεχωριστή νομική πράξη και θα ε, ε, ευχόμουν η Κομισιόν να μπορεί να μας ε, υποβάλει σχετικό χρονοδιάγραμμα. Αυτό έχει να κάνει με την προστασία των ζώων και φυτών, των άλλων ζώων των οργανισμών δηλαδή. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ξεχωριστή βάση για το θέμα αυτό. Θα χαιρόμουν αν μπορούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τώρα ήταν ε, αρνητικές οι εμπειρίες μου. Το 2007 μου είχαν υποσχεθεί ότι μέσα σε 12 μήνες ε, θα έχουμε σχετική πρόταση ε, σχετικά με την προστασία ζώντων οργανισμών. Έχουν περάσει 12 μήνες από τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσλέπω στην καλή συζήτηση. Παρακαλώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική οδηγία. Προφανώς και είναι τεχνική, αλλά βασίζεται ε, στην προστασία ε, και συγκεντρώνει έχουμε ε, άλλων οδηγιών όπως η 96 που θέτει πρότυπα ασφάλειας κατά της ε, Ιωνίζους Ακτινοβουλίας. Και βλέπετε, θα δείτε και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί, αλλά έχουμε και τις οδηγίες για τους ε, ασθενείς, για την πληροφόρηση σε περίπτωση ατυχήματος ε, και στους εργαζομένους εκτός του πυρηνικού τομέα. Νομίζω ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτή σε όλες αυτές τις οδηγίες. Το πρώτο ζήτημα είναι πάντα η αλλαγή της νομικής βάσης. Είναι μια οδηγία που βασίζεται στην ε, συνθήκη της Ευρατόμ. Όμως ο βασικός και κύριος στόχος αυτής της συνθήκης είναι η πυρηνική ανάπτυξη που θα διασφαλίσει την ευημερία και την ε, ειρήνη. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Η ε, ραδιολογική προστασία έχει τεθεί σε ισχύ για να προστατεύσει αυτή την ε, ε, πυρονική ασφάλεια. <coughs> Δεν είναι η περιβαλλοντική ασφάλεια ασφάλεια των καταναλωτών ή των ε, πολιτών. Δεύτερο επιχείρημα για την αλλαγή της νομικής βάσης είναι ότι εμείς ως ευρωβουλευτές πρέπει να έχουμε τη συναπόφαση ενώ αν πάμε στο πλαίσιο της συνθήκη Ευρατόμ, δίνουμε μόνο μια γνωμοδότηση. Εντελώς διαφορετικές λοιπόν οι δύο υποθέσει. Δεύτερο στοιχείο για αυτή την οδηγία. Ε, θέτει ένα ε, μεμονωμένο όριο δόσης ε, ενός μιλισιμπέρ ανά μονάδα πληθυσμού. Το ίδιο σε σχέση με την οδηγία 96. Όμως, αυτός ο αριθμός με όλα τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε, με τα όσα συνέβησαν στο Τσερνομπίλ, με όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μα για την εσωτερική μόλυνση, θα μπορούσαμε να το μειώσουμε από το ένα ε, μιλισιβέρτ να πάμε σε κάτι πολύ μικρότερο. Ε, ωστόσο, επιστώ την προσοχή στο γεγονό ότι σε αυτή την ε, οδηγία έχουμε εγκαταλείψει την συλλογική δόση. Δηλαδή, δεν λαμβάνουμε πλέον υπόψη τον αριθμό του ε, ατόμων που έχουν εκτεθεί σε σχέση με το επίπεδο της δόσης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί σημαίνει ότι αν αύριο ε, αφοπλίσουμε τα πυρηνικά εργοστάσια και εισαγάγουμε την απελευθέρωση, δηλαδή σε ένα επίπεδο θα μπορούσε να αποδεσμευθεί μια ε, ποσότητα ραδιενέργειας ε, που σέβεται τα επίπεδα δραστηριότητας ή συγκέντρωσης. Εκεί δεν λαμβάνουμε υπόψη την, ε, τον αριθμό των ατόμων που θα εκτεθούν. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και σοβαρό. Κάτι άλλο που υπάρχει είναι η αναφορά δόσης. Δηλαδή σε περίπτωση ατυχήματος κάθε χώρα μπορεί να πάει από τα 20 έως τα 50 μιλισιβέρ. Είναι μια τεράστια δόση. Μετά υπάρχει και μια φάση μετά το ατύχημα από τα 1 έως τα 20. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Φουκουσίμα. Εγώ πήγα εκεί και είπαν ότι έχετε δικαίωμα να πάτε μέχρι τους 20, μέχρι τα 20 μιλισιβέρτ και για τα παιδιά και τους ενήλικες για όλους. Είναι τεράστια ως δόση. Εκεί λοιπόν αποδεχόμαστε την ε, μόλυνση από τη ραδιενέργεια του, του περιβάλλοντος. Είναι εξαιρετικά σοβαρό Πρέπει να δούμε λοιπόν τι λέει και ο συνάδελφο εδώ πέρα σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Επίση για την προστασία των εργαζομένων. Από, τα 16, από 16 μέχρι 18 ετών μπορούν να πάνε μέχρι τα 6 μιλισιβέρτ ε, κατά έτο. Λε και αυτή η δόση είναι κάτι το αποδεκτό. Ή ότι δεν έχει κίνδυνο. Αν θέλετε, αυτή είναι μια αρνητική πτυχή της οδηγία σε σχέση με αυτά που είχαμε μέχρι τώρα. Και τελευταίο στοιχείο, που είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα μας ε, τα μέσα, είναι ότι αφορά την φιλελευθερωποίηση. Ε, γιατί μετά η αποδέσμευση και αποδοχή είναι μετά ο κανόνας. Στη Γαλλία δεν λέμε για παράδειγμα ότι απαγορεύεται. Και λέμε ότι απαγορεύεται και αν υπάρχει αδειοδότηση είναι κάτι ε, το προσωρινό. Είναι εξαιρετικά σοβαρό λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, ο Μύρος Ουσιασκή. Ε, e, e. Ευχαριστώ, πολύ σύντομα. Σε αντίθεση με τη συνάδελφο, εγώ συμφωνώ απολύτως με τον εισηγήτη. Δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη για την ε, Επιτροπή μας μπορεί να γίνει αποδεκτή για να αυξήσουμε το επίπεδο προστασίας ε, των πολιτών μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμεθα λοιπόν εδώ. Συμφωνούμε επίσης και με το γεγονός ότι μιλάμε για προστασία των ανθρώπων, αλλά και όλα αυτά που αφορούν ε, το περιβάλλον, τα ζώα κτλ. δεν έχουν θέση εδώ αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει ίσως κάποια κάπου ε, να υπάρξει μια διαβούλευση με τα μετρολογικά Ινστιτούτα και ούτω καθεξής να, να αναφέρεται λοιπόν κάτι τέτοιο κάπου, αλλά δεν αλλάζει κάτι στο χαρακτήρα της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ και θα σύντομα να δώσω το λόγο και στην Κομισιόν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, καλή και ισορροπημένη ε, έκθεση αυτή, καθώς και για τις επικοδομητικές τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν. Θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή είναι σημαντικό βήμα ε, για την προστασία από την ακτινοβολία. Πιστεύουμε ότι με το βήμα αυτό βελτιώνουμε σημαντικά την προστασία ε, των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Να απαντήσω σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Ο εισηγητής επί της αρχής επικροτεί την συμπερίληψη το, της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά θεωρεί ότι δεν υπάρχει ακόμα επαρκής επιστημονική βάση για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Κομισιόν πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα να συμπεριλάβουμε την προστασία του περιβάλλοντος στο παρόν σύστημα προστασίας ε, ανθρώπων και νομίζουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ε, με συνέπεια μόνο ε, στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom. Η ICEP έχει αναπτύξει ένα σύστημα Η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας, δηλαδή έχει ετοιμάσει ένα σύστημα ε, ε, για, την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Η σχετική έκθεση θα δημοσιευτεί σύντομα και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος κατά της Ακνοπολία. Σας Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή κυρία Ούλμερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι την επόμενη Τετάρτη από τις 3 ε, μέχρι τις 6.30 θα έχουμε ένα εργαστήριο για το θέμα αυτό. Ε, είσαστε προσκεκλημένοι. Θα χαρώ πολύ για την ε, συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την σύντομη παρέμβασή σα Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 5 Φεβρουαρίου, 20-21 Μαρτίου θα συζητήσουμε τι τροπολογίε. Ε, θα έχουμε συζήτηση στην Επιτροπή και 24 Απριλίου θα γίνει ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια. Θα γίνει η συζήτηση και η ψηφοφορία τον Ιούνιο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ε, σύντομη συζήτηση αυτή και ορίζω θέρμα τον ε, Υπουργό Υγείας της ε, Ιρλανδίας, ε, τον James Ράιλι. Καλώς ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είμαστε η μεγαλύτερη νομοθετική επιτροπή του Κοινοβουλίου, παρότι σήμερα συνεδριάζουμε σε μικρή αίθουσα. Ασχολούμαστε με πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει η οδηγία ε, για τον καπνό, οι διασυνοριακές απειλές προς την υγεία, το πρόγραμμα υγείας, ε, οι ιατρικές ε, συσκευές, τα ιατρικά βοηθήματα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθείτε κι εσείς και περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίασή σας. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά και κατόπιν θα ακούσουμε τους συντονιστές και σε έναν δεύτερο γύρο θα μπορέσουν οι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Μία εισηγήτρια ήδη ζητάει το λόγο. Έχουμε πάρα πολλούς εισηγητές μαζί μας εδώ σήμερα. Ε, θα είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Κύριε Ράιλε, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρίας στην τομέα της υγεία. Το 2013 ε, γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την ε, προσχώρηση της Ιρλανδία ε, στην, στην ΕΟΚ. Για μας που ήμασταν ε, και τότε το 1973 και συμμετείχαμε είναι τρομερές επιτυχίες που είχαμε στο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη. Από τότε που ε, προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αμέτρητα τα ωφέλη για τους Ελληναδούς ε, πολίτες και ε, από οικονομικής και από κοινωνικής σκοπιάς. Ωστόσο υπάρχουν διάφορες προκλήσεις τώρα, δεδομένες και της οικονομικής κατάστασης. Γι' αυτό τον λόγο το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας έχει ως στόχο να κάνει προτάσεις που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Ευρώπης, δηλαδή σταθερότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Παρά λοιπόν την οικονομική κατάσταση, παλεύουμε για να βελτιώσουμε την υγεία και ευημερία των πολιτών μας, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν συστήματα που στηρίζουν και βελτιώνουν την αποδοτικότητα ε, σε ό,τι φορά την υγειονομική περίθαρψη και τους πολίτες μας. Και κάθε, ενώ κάθε κράτος μέλος αντιμετωπίζει τη δική του πραγματικότητα στον τομέα της υγείας, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία ε, και ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του Κοινοβουλίου είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Ε, είστε άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ο ρόλος σας ως ε, συνομοθετών είναι κρίσιμη σημασία για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους. Η Ιρλανδική Προεδρία αναγνωρίζει τη σημασία συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο με το να συνεργαστούμε μαζί σας ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις ε, ζωές των πολιτών μας τώρα αλλά και στο μέλλον. Μαζί μας ε, έχουμε και, την, και το τρίο της Προεδρίας, η Λιθουανία και η Ελλάδα και βεβαίως προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία με τους συναδέλφους και με τον δόκτορα Κάτης η Ιρλανδική Προεδρία θα αξιοποιήσει τους πόρους της ε, για να θέσει προτεραιότητες και να σημειώσει σημαντική πρόοδο σε μια σειρά βασικών νομοθετικών ε, φακέλων για την υγεία, όπως είναι τα προϊόντα καπνού, διασυνορικές απειλές για την υγεία, κλινικές δοκιμές, ε, η, ανάπτυξη, υγεία για την ανάπτυξη και ιατρικός εξοπλισμός. Το κάπνισμα πρώτα απ' όλα είναι από τις μεγαλύτερες απειλές ε, ε, για τη δημόσια υγεία και περίπου 700.000 Ευρωπαίοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Εκατομμύρια ακόμα ε, αναγκάζονται να ζήσουν με το βάρο ε, χρόνιων ασθενειών που προκαλούνται από την κατανάλωση καπνού. Το κόστος ε, για τα μεμονωμένα άτομα αλλά και τι οικογένειε τους ό,τι αφορά την απώλεια υγιών ε, χρόνων ζωής, η απώλεια μελών της οικογένειας και ε, όλα τα βάσανα που προκαλούνται είναι πραγματικά ανυπολόγιστα. Και η μεγάλη τραγωδία εδώ είναι ότι είναι κάτι που μπορεί να αποφευθεί. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν. Να βοηθήσουμε του καπνιστέ να σταματήσουν το κάπνισμα και να αποτρέψουμε του νέου να το ξεκινήσουν. Ε, πέραν του ανθρωπίνου κόστος υπάρχει και ένα ε, τεράστιο οικονομικό κόστος γιατί η θεραπεία των ασθενών και η περίθαλψή τους ε, έχει ένα πραγματικά ογκοδέστατο κόστος. Η κατανάλωση ε, προϊόντων καπνού όμως έχει και ευρύτερες ε, αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, απουσία από το χώρο εργασίας, απώλεια σε παραγωγικότητα και προώρηση δεξιοδότηση. Η νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα είναι βασική προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία. Ε, ιδίω σε ό,τι φορά και τα παιδιά. Στην Ιρλανδία βλέπουμε ότι το 78% των ε, καπνιστών ξεκινούν το κάπνισμα πριν από την ηλικία των 18. Ε, όταν ακόμα είναι παιδιά δηλαδή. Και βεβαίω όταν κάποιο ξεκινά το κάπνισμα είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσει μετά από χρόνια, μπορεί και ποτέ. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στο τέλος ένας στους δύο καπνιστές θα χάσει τη ζωή του από μία ασθένεια που συνδέεται με το κάπνισμα και αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι τα μέτρα ελέγχου του καπνού ε, που λαμβάνονται σήμερα ε, δεν ε, προστατεύουν μία από τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία του ε, ευρωπαϊκού πληθυσμού και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε ε, τον καπνιστή που σε τελική ανάλυση είναι και Ευρωπαίος πολίτης. Η νομοθεσία αυτή είναι βασική προτεραιότητα λοιπόν για την δική μας Προεδρία και είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι μπορώ ε, για να σημειωθεί η περίοδος. Τον προηγούμενο Αύγουστο εγώ και άλλοι εννέα Υπουργοί Υγείας αποστήλαμε επιστολή προς την Επιτροπή για να ε, δημοσιευθεί η πρόταση μέχρι το τέλος του 2012 και χάρηκα που η Επιτροπή την ε, δημοσίευσε στις 19 Δεκεμβρίου. Ξέρω ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες. Ε, στο παρελθόν η βιομηχανία έχει αποδείξει πως η μεγάλη επίδραση μπορεί να έχει και ότι θα αξιοποιήσει σε οποιοδήποτε μέσο για να ασκήσει πιέσεις ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την νομοθεσία. Θεωρώ ότι εμείς ως νομοθέτες, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, πρέπει να θέσουμε τα συμφέροντα των ε, πολιτών μας ε, πάνω απ' όλα και να εργαστούμε για την ε, έγκαιρη υιοθέτηση της νομοθεσίας. Στον επόμενο μήνα θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για αυτό το ζήτημα. Προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής σας, αλλά και ιδίως με, με την Λίντα Μακάβιν, που μόλις ορίστηκε ως εισηγήτρια για να διασφαλίσουμε ότι θα υιοθετηθεί αυτό το, αυτή η νομική πράξη στο στομότερο δυνατόν. Στο ευρύτερο θέμα της, ε, του ελέγχου καπνιστού, του καπνού ήμασταν πρωτοπόροι σε ό,τι αφορά την ε, ε, προστασία των εργαζομένων και της υγείας τους με την υιοθέτηση απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους εργασίας. Το Μάρτιο, κατά το Συμβούλιο, θα εξετάσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τι πρέπει να γίνει ακόμα για να ε, διασφαλίσουμε ένα ασφαλές άκαπνο περιβάλλον σε όλους τους πολίτες. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, είμαστε ειλικρινεί. Αν αυτό το προϊόν ε, ε, βρισκόταν στην αγορά ε, ή μάλλον έμπαινε στην αγορά αυτή τη στιγμή γνωρίζοντα τα όσα γνωρίζουμε, δεν θα το επιτρέπαμε. Από το 2014 μέχρι το ε, θα έχουμε ένα νέο ε, πρόγραμμα ε, υγείας, το οποίο βασίζεται σε αυτό που λύγει φέτος. Σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα θα εστιαστούμε σε έναν μικρότερο αριθμό συγκεκριμένων στοχευμένων δράσεων με προστιθέμενη εξήγηση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γενική στόχη είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της περίθαλψης αλλά και της βιωσιμότητας των υγειονομικών μας συστημάτων για να αυξήσουμε να βελτιώσουμε την υγεία των πολιτών μα και να του προστατεύσουμε από τις διασυνεριακέ απειλές. Ε, χαιρετίζω τι προόδου που έχουν σημειωθεί διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Ωστόσο, υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Δύο από αυτά έχουν οριζόντιο χαρακτήρα. Ο προπολογισμό του προγράμματο και το ζήτημα των καταξιδότηση και εκτελεστικών πράξεων για τα ετήσια προγράμματα εργασιών. Άλλο ζήτημα είναι ο μηχανισμό χρηματοδότηση για τι κοινέ ε, δράσει. Η Ιλλανδική Προεδρία ε, ε, είναι απολύτως ετεθειμένη να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσει και να εργαστεί επικοδηματικά μαζί με το Συμβούλιο, θα, με το Κοινοβούλιο. Ε, θα βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία και με την κυρία ε, εισηγήτρια. Ε, Βεβαίω ε, θα επηρεαστεί το έργο μα και από τι διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ελπίζουμε να υπάρχουμε αρκετό χρόνο για την υλοποίηση του προγράμματος από τις αρχές 2014. Πρόσφατα έχουμε δει μεγάλο αριθμό διασυνοριακών απειλών, όπως ο ΙΤΑ 1 η 1, η ε, γρήβη των πτυνών και το καθεξής. Είδαμε βέβαια ότι ο αντίκτυπος αυτών των πανδημιών δεν ήταν ε, όσο, αναμε... όσο μεγάλος όσο αναμενόταν, όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να είμαστε σίγουροι ότι όλοι οι πολίτες μας θα έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό και βεβαίω η διασυνορική συνεργασία είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη. Η Ιλλανδική Προεδρία είναι διατεθειμένη να, να διαπραγματευτεί με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία και πάλι με ε, ε, ε, τον εισηγητή Πανιού. Θα έχουμε έτσι μια νομική βάση για την κοινή προμήθεια εμβολίων και για την λήψη άλλων μέτρων για την προστασία των πολιτών από τέτοιες πανδημίες. Η απόφαση θα πρέπει επίσης ε, να τονίσει τη σημασία ε, της ε, συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Οι τριμερείς διάλογοι με το Κοινοβούλιο θα ξεκινήσουν στις επόμενες εβδομάδες. Πολλά μένουν να συζητηθούν για την εξουσιοδότηση της Επιτροπής, για τη λήψη αποφάσεων, για την ετοιμότητα και τα προγράμματα πρόληψης. Είμαστε τεθειμένοι είμαστε σίγουροι ότι μπορούν αυτά να επιληθούν με ένα επαγγελματικό πνεύμα συνεργασία το συντομότερο δυνατόν. Και έτσι βασιζόμαστε στη δική σα συνεργασία ω προ αυτό, αλλά και στη συνεργασία τη Επιτροπή. Για τις κλινικές δοκιμές η πρόσβαση ε, σε νέα καινοτόμα φάρμακα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους ε, πολίτες μας. Οι κλινικές δοκιμές είναι απαραίτητες για να ε, επιτρέπουν την πρόσβαση σε τέτοια φάρμακα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των σκευασμάτων. Ιδίω ό,τι αφορά τα, τα, τα σκευάσματα για ανθρώπινη χρήση που έχουν ως στόχο την ε, βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Είναι πολύ σημαντικό και για τον ε, τομέα της φαρμακοβιομηχανίας. Είναι τεράστιο και το διοικητικό άκθος αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν, υπάρχει σημαντική πρόοδος. Θα συναντηθώ με την εισηγήτρια Γκάλνης Βίμαρκ ε, στη συνέχεια. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η πρόταση και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει έγκαιρη συμφωνία. Θέλουμε να υπάρξει πρόταση και για τον ιατρικό εξοπλισμό βάσει της πρότασης ε, του Σεπτεμβρίου του 2012. Στόχος είναι ε, να υπάρξει ένα βελτιωμένο νομικό ε, πλαίσιο για τον ιατρικό αυτοεξοπλισμό και τον in vitro διαγνωστικό εξοπλισμό. Κατανοώ τις, ε, τον προβληματισμό των πολιτών και, το, και πολιτικών ε, μετά το σκάνδαλο με τα επιτέρματα σιλικόνης. πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα και τα σκευάσματα για τους πολίτες μας. Όμως παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και η βιομηχανία, ο κλάδος ε, παρέχει ασφαλή προϊόντα με έγκαιρο τρόπο προς όφελος ε, των ε, πολιτών. Οι βελτιώσει στην ιατρική τεχνολογία μπορούν να αυξήσουν και την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσουν θέσει εργασία, μειώνοντα το κόστο υγειονομική περίθαλψη και τη βελτίωση τη ποιότητα και τη αποτελεσματικότητα τη περίθαλψη. ε, προτείνεται προτείνονται γενικότερη αξιολόγηση και πριν από τη θέση σε εμπορία. Είναι περίπλοκες οι προτάσεις, όμως είναι δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος κατά τη διάρκεια της Ιλλανδικής Προεδρίας. Ε, συνάντησα και την εισηγήτρια χθε, αλλά και την ε, σκιώδη εισηγήτρια και θα συναντήσω τον εισηγητή για την πρόταση in vitro στη συνέχεια. Η Ιρλανδική Προεδρία παρακολουθεί ε, και τις συζητήσεις ε, για άλλες οδηγίες, ε, ιδίω ό,τι αφορά την οδηγία, την οδηγία περί διαφάνειας και χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας σε αυτή την ε, Επιτροπή. Έχουμε σημειώσει την ε, διστακτικότητα κάποιων μελών να συνεχιστεί η εξέταση της πρότασης. Η Προεδρία μπορεί να εισέλθει στις διαπραγματεύσεις με άλλα ε, θεσμικά όργανα μόνο αν υπάρχει ε, ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Ε, προτίθεμαι να διαρευνήσω αν υπάρχει στήριξη από το Συμβούλιο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ξεκινώντας από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του επόμενου μήνα για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα. Τώρα, να αναφερθώ σε κάποια άλλα ζητήματα του προγράμματο. Ε, σε ό,τι φορά την σημασία τη έρευνα και καινοτομία, η Προεδρία ε, θα διοργανώσει μία. Ένα συνέδριο, μια συνδιάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ηλεκτρονική υγεία, αλλά και μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομία και Έρευνα, μια συνδιάσκεψη για το μέλλον τη ε, ε, της έρευνας σε ό,τι αφορά τον εγκέφαλο. Ε, για την ηλεκτρονική υγεία θα λάβει χώρα στις 13 15 Μαΐου. Και φέτος το βασικό θέμα θα είναι η ηλεκτρονική υγεία και η καινοτομία σε ό,τι αφορά την ευημερία. Η δεύτερη συνδιάσκεψη θα είναι συνδιάσκεψη εμπειρογνώμων υψηλού επίπεδου. Ε, θα συνδιοργανωθεί με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Καινοτομία και θα λάβει χώρα στις 27 και 28 Μαΐου 2013 ε, για να προστιμήν και του Ευρωπαϊκού Μήνα Εγκεφάλου. Έχουμε και μια άτυπη συνάντηση με τους Υπουργούς Υγείας στις 4 και 5 Μαρτίου στο Δουβλίνο ε, με βασικά ζητήματα την υγεία και ευημερία. Θα έχουμε θέματα και για το άκαπνο περιβάλλον, την ασφάλεια των ασθενών, και τα παιδιά με, με πολύπλοκες αναπτυξιακές ανάγκες συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σα. Ε, εκτιμώ ιδίω αυτή τη ε, ε, δυνατότητα που μου δώσατε να σα ενημερώσω για τι προτεραιότητε τη Ισλανδική Προεδρία στην τομέα τη υγεία και να απαντήσω βεβαίω και στι ερωτήσει σα. Όπω είπα, έχουμε θέσει προτεραιότητε στην ατζέντα μα και πιστεύω ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσουμε του πόρου μα. Ε, το εύρο των μέτρων ε, που εμεί ω ε, συνομοθέτε έχουμε στη διάθεσή μα είναι εξαιρετικά σημαντικά και για την υγεία των πολιτών και για τη στήριξη τη καινοτομία και έρευνα στην Ευρώπη. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σα με επικοδομητικό τρόπο για να προαγάγουμε την ατζέντα τη υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα να ανοίξουμε το γύρο τώρα των πρώτων ερωτήσεων. Ε, συνηθίζεται σε εμά να ξεκινούν οι ε, ε και το, ε, το, πρώτο το λόγο έχει ο Πίτερ Λίζε που είναι συντονιστή ε, του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα, Σα ευχαριστούμε για την εισαγωγή σα. Ε, αναφερθήκατε στα προϊόντα καπνού ήδη στην αρχή της παρεμβασή σα. Σας ε, ευχαριστώ που δεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μας ε, να συμμετάσχετε σε ακρόαση. Είναι πρόταση του ΕΛΚ και χαίρομαι που εσείς ως προεδρεύων και μάλιστα από κόμμα που ανήκει στο ΕΛΚ θα συμμετάσχετε. Θα γίνουν πολλές συζητήσεις σχετικά με την οδηγία για τον καπνό αλλά ε, σε ένα θέμα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα του παθητικού καπνίσματος ε, και του κινδύνους για τα παιδιά ιδιαίτερα. Τα μηνύματα, τα προειδοποιητικά που λαμβάνουμε κυρίως έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον καπνιστή, αλλά θα πρέπει ε, να γνωρίζουμε ότι ε, τα παιδιά και ιδιαίτερα τα βρέφη εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους. Αναφέρεται ο ξαφνικός θάνατος ε, παιδιών και συνδέεται με το κάπνισμα σύμφωνα με κάποιες μελέτες. Δεύτερον, Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν εμπίπτει άμεσα στι αρμοδιότητέ σα, ε, έχει να κάνει όμω ε, με την υγεία των ανθρώπων και πρόκειται για την οδηγία αναγνώριση ε, των επαγγελματικών προσόντων. Η Επιτροπή μας είπε στην επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή ότι δεν Θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα που υπάρχει σε κάποια κράτη-μέλη ε, με δεκαετή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση να μπορεί κανείς να γίνει νοσοκόμος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό με τον αρμόδιο Υπουργό στο Συμβούλιο. και η ε, ε, ε, αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς είπε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα της ε, δεκαετίας, ε, της δεκατούς ε, πρακτικής άσκησης, η εκπαίδευση δεν ξεκινάει με το, με το πολιτήριο λυκείου. Πολύ συχνά οι νοσοκόμες που έχουν δεκαετή κατάρτιση γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα που είμαι γιατρός. Η Λίντα Μακέιβαν, να δώσω το λόγο στη συνάδελφα πρώτα που πρέπει να φύγει. Χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Όπως γνωρίζετε Έχω πολύ ισχυρέ απόψει όσον αφορά τον καπνό και ξέρω ότι συμφωνείτε μαζί μου, αλλά θα ήθελα να, διαβεβαιώσετε, να μας διαβεβαιώσετε ότι θα θυμίσετε σε όλους τους συναδέρφους σας στο Συμβούλιο ε, ε, ε, αυτά που έχει πει ο ΠΟΗ ότι όπου είναι απαραίτητε οι συνδιαλλαγέ με την βιομηχανία καπνού θα πρέπει να είναι διαφανεί οι επαφέ. Ε, ξέρετε τι έχει γίνει με την σχετική βιομηχανία. Έχει προσπαθήσει παρασκηνιακά να ε, καθυστερήσει την ομοθεσία ε, και αυτό δεν πρέπει να γίνει με κανέναν τρόπο. Είμαι πεπισμένη ότι και εσείς έχετε ισχυρέ απόψει όσον αφορά την οδηγία για τον καπνό. Παρακαλώ να επηρεάσετε και τους ε, ε, συναδέλφους σας στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Γκροστέτ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Σας άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όλα τα συστήματα στα οποία αναφερθήκατε είναι εξαιρετικά σημαντικά για την Επιτροπή μας η συγγήτρια του τρίτου προγράμματος ε, δράσης στον τομέα της υγείας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αναφερθήκατε σε αυτό και μάλιστα διεξοδικά. Είπατε τι μένει ακόμα να γίνει και πράγματι είχαμε πολλές συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου ε, και εξετάσαμε ακόμα τρία στοιχεία, το επίπεδο της χρηματοδότησης, ε, και το καθεξής. Για τον τελικό ε, χρηματοοικονομικό φάκελο να σας ε, θυμίσω ότι για το κοινοβούλιο μας αυτό το ζήτημα είναι θεμελιώδου σημασία και αν δεν το λάβουμε δεν θα συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Θα σας υπενθυμίσω ότι η χρηματοοικονομική κατανομή είναι ήδη εξαιρετικά δύναμη. 146 ε, εκατομμύρια για την περίοδο 14-20. Παρά τα όσα γνωρίζουμε για τον προπολογισμό, τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν για την ε, συμφωνία, για τον προπολογισμό αυτών, δεν ε, μπορούμε να φανταστούμε πώς θα θυσιάσουμε και την κατανομή όπως έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εμφιστώ λοιπόν την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα, γιατί μιλάμε για πολλά διαφορετικά προγράμματα σε ό,τι αφορά ε, την ε, πάλι κατά των σπάνων ασθενειών, του αλκοόλ και του καθεξής. Και, όπως είπαμε και στην αρχή, ε, ε ένας πληθυσμός που βρίσκεται σε καλή υγεία έχει, καλύτερες, ε, και έχει πολλά ωφέλη και για την ε, παραγωγικότητα της οικονομίας. Να εφιστείτε την προσοχή σας και σε κάτι άλλο, ε, με το οποίο συμφωνώ μαζί σας, ε, δηλαδή σε ό,τι αφορά το φαρμακευτικό τομέα στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα που με απασχολεί πολύ, γιατί δύο φορές ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αδειοδότηση σε ένα ε, φάρμακο ε, κατά των σπάνιων ασθενειών, το μοναδικό φάρμακο, το οποίο όμως επιτίθεται στο ύπαρ και πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο, Δυο φορές λοιπόν υπήρξε αυτή η αδειοδότηση για να τεθεί σε εμπορία το φάρμακο αυτό που ε, χρησιμοποιείται εδώ και 20 χρόνια στην Ευρώπη και επανέρχεται η Επιτροπή σε, αυτό, σε αυτή την απόφαση. Ε, βασίζομαι σε εσά λοιπόν ε, για να ασκήσετε πιέσεις για να μην υπάρξουν ε, άλλοι ελιγμοί στην Επιτροπή σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ που τήρησα το χρόνο των δύο λεπτών. Η συνάδελφος Ροτ Πέρεντ για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που ε, βρίσκεστε πάλι εδώ. Ε, πολύ σύντομα. Πιστεύετε ότι όσον αφορά τα ιατρικά βοηθήματα τι ιατρικέ συσκευέ θα πρέπει ε, να κάνουμε κάποιε αλλαγέ. Ε, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ε, διάκριση ανάλογα με το είδο και ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι για μερικέ θα πρέπει να υπάρχει απλά κοινοποίηση, ενώ για άλλε θα πρέπει να υπάρχει έγκριση πριν τη χρήση του σε ασθενεί. Και αν συμφωνείτε μαζί μου, συμφωνείτε επίση ότι στι περιπτώσει κοινοποίηση θα πρέπει να ε, εξετάζουμε τους φορείς κοινοποίησης ε, και ε, τις απαιτήσεις για γνώσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν στις φορείς κοινοποίησης και συμφωνείτε επίσης μαζί μου ότι όσον αφορά την ταξινόμηση ή την, τον καθορισμό για, για μια χρήση πολλαπλέ ε, χρήσει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε του ε, κανόνε υγιεινή και άλλου ε, όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή των βοηθημάτων αυτών, αλλά να καθορίσουμε τι είναι μία χρήση, τι είναι οι πολλαπλές χρήσεις και πώς γίνεται και η σωστή απόρριψη των προϊόντων αυτών μετά τη χρήση τους. 31 δευτερόλεπτα ε, ε, χρωστάω στη Ροτ Μπέρεντ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ ε, εδώ. Ο Καρλ Έχω τρακ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω μία ερώτηση σχετικά με τον καπνό. Η Κομισιόν ασχολείται πολύ με το θέμα της ενιαίας συσκευασίας Και ακούω να λένε ότι η Κομισιόν ξεπερνάει εδώ τι αρμοδιότητε τη. Ε, σε τι βαθμό είναι αλήθεια αυτό, υπάρχει. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος να καταλήξουμε κάποτε στο δικαστήριο και να τεθούν ένα σωρό ερωτήσεις ε, για το λόγο αυτό. Ευχαριστώ πολύ και τέλος ο Γκλένις Βίλμετ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ, σας ε, καλωσορίζω. Ε, χαίρομαι που τον ε, κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές τον έχετε βάλει στην κορυφή του θεματολογίου σας ως εισηγήτρια για τον συγκεκριμένο κανονισμό και είμαι ευγνώμων για τη συνεργασία που ήδη είχαμε την ομάδα σας, αλλά το ένα θέμα που ανακύπτει για μένα είναι το θέμα της διαφάνειας αποτελεί ε, πραγματικό πρόβλημα η αξιοπιστία των κλινικών δοκιμών και συχνά οι ε, επιστήμονες δυσκολεύονται να, να ε, βρουν τα στοιχεία για να ελέγξουν τα αποτελέσματα των δοκιμών. Πολύ συχνά ξέρουμε ότι παρακρατούνται στοιχεία, δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία, οι κλινικές δοκιμές μπορεί να ε, γίνουν πολλές φορές ε, προτού να ε, γίνει γνωστό ότι είναι μια αποτελεσματικές ή επικίνδυνες. Δεν νομίζω όμως ότι ε, η πρόταση της Επιτροπής είναι αρκετά φιλόδοξη. Συμφωνείτε ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Άλλωστε, οι ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινικές ε, δοκιμές ε, θέλουν να προωθήσουν την γιατρική για τους ίδιους και για άλλους συμπάσχοντες, όχι για να ωφεληθεί μια συγκεκριμένη εταιρεία. Πιστεύω ότι η αξιοπιστία στη γιατρική αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών για τις θεραπείες αυτές θα αποτελέσει αποτέλεσμα τι μεγαλύτερε διαφάνειε στις κλινικές Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο. Σας παρακαλώ να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Σε πρώτο να προχωρήσουμε στο δεύτερο γύρο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, τους αγαπητούς ε, βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Θέλω να πω εξ αρχής ως μέλος του Συμβουλίου και ασκών την ε, Προεδρία, ε, βασικός μας γνώμονας είναι ο ασθενής. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, σημείο κίνησης, να απαντήσω σε αυτό που είπατε για το παθητικό κάπνισμα και για τα παιδιά. Συμφωνώ και εγώ ότι χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά σε αυτό το τομέα και να επισημαίνω ειδικά ότι τα παιδιά είναι μια ευάλωτη ομάδα. Είναι ανήλικοι, Άρα έχουμε το καθήκον να τα προστατεύσουμε ως κοινοβούλιο, ως κομισιόν, ως συμβούλιο. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά, στην ίδια παράταξη όλοι προκειμένου. Μόνο ακόμα και ο καπνιστής δεν θέλει να δει το παιδί του να καπνίσει. Ακόμα και ο ίδιος ο καπνιστής. Άρα η γονική συμπεριφορά είναι πολύ σημαντική. Τα παιδιά δεν είναι ανόητα ακούν τι τους λένε, αλλά βλέπουν κιόλα τι κάνουν οι μεγάλοι. Άρα το να το λες από τη μία πλευρά το κάπνισμα κάνει κακό, σου μικράνει τη ζωή, θα σου δημιουργήσει προβλήματα υγείας, αρτηριακές, καρδιακές νόσους, έμφραγμα κτλ. Πέστε αυτά. Αλλά όταν βλέπουν το γονιό που τον σέβονται και τον εμπιστεύονται, τη μάνα, τον πατέρα, τους βλέπουν να κάθονται και να καπνίζουν ένα τσιγάρο, ό,τι και να πεις, δεν έχει νόημα. Άρα πρέπει να γίνει δουλειά στην ανατροφή των παιδιών και να βοηθήσουν τους γονείς να βρουν τον κατάλληλο τρόπο να προστατεύσουν τα παιδιά τους από μια πολύ κακή συνήθεια που σκοτώνει έναν στους δύο καπνιστές. Αυτά τα δεδομένα. Ό,τι και να λέμε δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Οπότε δέχομαι αυτό που είπατε για την εκπαίδευση των κηδεμόνων και θα το λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά τώρα την διαφάνεια σε συναντήσεις με τη την καπνοβιομηχανία, πράγματι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Και θέλω να καταγραφεί και η ευγνωμοσύνη μου για τη δική σας ε, υποστήριξη προκειμένου. Έπειτα είπατε και κάποια λόγια για τον προπολογισμό και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει αλλά δυστυχώ ούτε είναι κάτι που ελέγχω, ούτε είναι στην αρμοδιότητά μου. Φυσικά και θα δώσουμε μάχη για τον προπολογισμό. Αν ε, εξαρτώνταν από μένα, εγώ τον άφησα τον προπολογισμό. Η υγεία είναι ο πλούτο μα, δηλαδή τι να είσαι πλούσιο, αν είσαι άρρωστο και δεν μπορούσε να το ε, χαρίσει να χαρίσει τη ζωή σου. Γι' αυτό δεν λέμε κιόλα ότι είναι καλύτερα να έχει την υγειά σου παρά να έχει λεφτά, να είσαι πλούσιο. Τώρα, για να βοηθήσουμε τους αγρότες να παραμείνουν στην ε, Ευρώπη, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνουν και οι κλικές δοκιμές. Αλλά θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή. Όλα αυτά γίνονται χάρη των ασθενών. Άρα οι κλινικές δοκιμές γίνονται για την καλύτερη προστασία των ασθενών. Άρα η διαφάνεια, τα δεδομένα, τα στατιστικά στοιχεία είναι όλα κρίσιμες σημασία. Αν τώρα η όλη ιατρική βιομηχανία ιατρικού εξοπλισμού δείχνει μια κάποια α, μυστικοπάθεια, αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε καν την ίδια. Για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, ε, πράγματι είχαμε μια χθεσινή συνάντηση και τα συζητήσαμε κιόλα και διμερώς. Σα ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στην εναρμόνιση των φορέων κοινοποίηση στην Ευρώπη. Και τα πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούν φυσικά και αυτό θα είναι πρόκληση για κάποιε χώρε, Αλλά πιστεύω ότι αν ξεκινώντα έχοντα ω σημείο κίνηση το συμφέρον των ασθενών είμαστε στην κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες της επανεπεξεργασίας, συμφωνώ. Πρέπει να ορίσουμε ποια είναι τα προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, με την, ε, τα κατάλληλα πρότυπα υγιεινής στα νοσοκομεία και ποια είναι τα άλλα νοσοκομιακά υλικά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. η ομοιομορφία και η εναρμόνιση των προτύπων είναι κρίσιμη σημασία για όλους τους πολίτες μας. Κύριε Φλόρανς, σε ό,τι αφορά ε, το γεγονό ότι η Κομισιόν ξεπερνά τα εσκαμμένα, κοιτάξτε, ό,τι και να με εμεί, δεν ξέρουμε πώ θα αντιδράσει η βιομηχανία. Α δούμε το παράδειγμα τη Αυστραλία, εμείς πρέπει να ε, κρατήσουμε το στόχο μας, να έχουμε μια οδηγία των στομάτων δυνατών. Ξέρετε, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι προφανές. Συχνά δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε την αιτία των προβλημάτων. Ο καρκίνο ε, είναι ένα τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, γνωρίζουμε πολλά για τον καρκίνο, αλλά χρειάζεται να μάθουμε πολλά περισσότερα, να καλύψουμε πολλά περισσότερα. Όταν όμω γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα, τι προκαλεί τον καρκίνο, όταν, όταν τελικά βρούμε την αιτία του καρκίνου, θα πρέπει να κινηθούμε άμεσα για να αντιμετωπίσουμε την αιτία τώρα. Οι καπνιστές, όσοι επιθυμούν να καπνίζουν, ε, κοιτάξτε, δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του είναι να καπνίζουν, δεν μπορούμε να του απαγορεύσουμε, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή ε, των παιδιών, των ανήλικων και όσων ε, βρίσκονται στο περιβάλλον του. Κύριε Πρόεδρε, ω Ιρλανδό, ε, αυτό το θέμα ε, του καπνίσματος, του παθικού καπνίσματος των παιδιών ε, που εισπραίνουν τον καπνό των γονέων στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου είναι κάτι που με σοκάρει. Για τη διαφάνεια, όπως είπα και πριν, συμφωνώ και επαυξάνω στο παρελθόν. Ξέρετε, ως γιατρός μιλάω. Όταν ε, ένα νέο τολικό φάρμακο στις δοκιμές φάνηκε πολύ αποτελεσματικό, ήταν πολύ καλό. Αλλά ταυτόχρονα φάνηκαν αποτελέσματα κατά καρδιοπαθών, τα οποία δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ. Αυτό είναι πραγματικά ε, τραγικό. Πρέπει να προστατεύουμε τους πολίτες μας. Και σίγουρα η βιομηχανία όταν κινείται έτσι δεν εξυπηρετεί ούτε δικά τη συμφέροντα, γιατί δεν είναι προ όφελό της ε, να υπάρχει τέτοια έλλειψη εμπιστοσύνη. Καθώς η ε, ασθενείς ε, καταναλώνουν τα φάρμακα με καλή την πίστη και οι γιατροί ε, συνταγραφούν τα φάρμακα καλή την πίστη. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι όσο μπορούμε, αλλά όπως λέω και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει, θα πρέπει να παντρέψουμε την ανάγκη για γρήγορη δράση με την ρεαλιστικότητα και την αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει δηλαδή πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές απειλές για την υγεία των Ευρωπαϊκών πολιτών μας, οπότε αυτό θα το κάνουμε με την πρόθεση της οδηγίας. Περιμένω τη δική σας υποστήριξη και εγώ μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου. Φτάνουμε στο δεύτερο γύρο. Και θα δώσω την δυνατότητα στον Καλχάνς Φλόρενς να θέσει συμπληρωματική ερώτηση, δεν απαντήθηκε η ερώτησή του. Ε, πρώτα όμως, η Μιζέλ Δεν είναι πια παρούσα. Αχ, instead of Karl Schlüter. Ο Καρλ Σλούτερ. Λίντα Μακέβαν. Λίντα Μακέβαν. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα στην ε, Επιτροπή μας και χαίρομαι που είναι εδώ και ο Υπουργό Υγείας της Λιθουανίας εδώ σήμερα, διότι ε, θα έχουμε τρεις ε, σημαντικές νομοθετικές προτάσεις για την υγεία τους επόμενους μήνες και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να σημειώσουμε πρόοδο. Ορίστηκα εισηγήτρια για την οδηγία του καπνού και εσείς είπατε ότι θέλετε πρώτα να θέσετε τα θέματα υγείας. Συμφωνώ απόλυτα. Θα υποβάλω προτάσεις ε, να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν και να φροντίσουμε να έχουμε μια, έναν καλό κανονισμό για τη βιομηχανία καπνού. Δεν ε, έχουμε αρχίσει τις ε, συζητήσεις εντός του Κοινοβουλίου ακόμα, δεν ξέρω καν ποιοι είναι οι σκιώδες αλλά όλες οι πολιτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου εργάστηκαν σκληρά ε, πριν τα Χριστούγεννα για να τεθεί επιτάπητο στο θέμα αυτό. Πιέσαμε την ε, Επιτροπή διότι ε, φοβηθήκαμε ότι δεν θα προλάβει η παρούσα θητεία αλλά τώρα έχουμε την πρόταση και κοιτώ όλου του συναδέλφου. θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην οδηγία για τον καπνό. Το χρωστάμε αυτού του πολίτε μα. Ο Πέτερ Λίζε αναφέρθηκε σε ένα θέμα. Ε, ε, διαπιστώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός ε, των παιδιών με άσθμα μετά την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Πριν είχαμε ποσοστό 12%, τώρα έχουμε 2% παιδιών με άσθμα. Στην ε, Σκοτία είδαμε πτώσεις ε, στις καρδιακές παθήσεις από τότε που ξεκίνησε η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, κάτι που έχει οδηγήσει και σε μεγάλη πτώση του αριθμού των καπνιστών στις χώρες αυτές. Ε, είναι κάτι λοιπόν που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνω. Ελπίζω στην υποστήριξή σας. Υπάρχει και ε, ε, ε, μια άλλη αιτία θανάτου η οποία μπορεί να αποφευθεί. Δεν ξέρω αν είδατε στην είσοδο υπάρχει μια έκθεση σχετικά με το μονοξίδιο του άνθρακα. Κάποιοι συνάδελφοί μου νομίζω ότι θα σοκαριστούν αν δουν τον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν από δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα στις χώρες τους. Πέρσι στη Γερμανία 10 άνθρωποι πέθαναν λόγω χρήσης γκριλ και αλλού υπάρχουν πολλοί θάνατοι από, διοξίδιο, από συγγνώμη, μονοξίδιο του άνθρακα. Ε, υπάρχουν οι ανιχνευτές ε, μονοξιδίου του άνθρακα. Ε, θα πρέπει ε, να γίνεται καλύτερα επισήμανση στα γκριλ στις ψηστιέρες δηλαδή. Ε, επίσης ε, ε, έχουμε δει ε, σε, ξενοδοχεία στην Ευρώπη, έχουμε θανάτους από μορφή του άνθρακα. Δύο παιδιά από την εκλογική μου περιφέρεια πέθαναν στην Ελλάδα από δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος Μπόρς, και μάλιστα σε πολλού τομεί. Πάντω είναι σημαντικό θέμα τη δημόσια υγεία και μπορούμε να αποφύγουμε θανάτου από την αιτία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λίντα Μακέβαν. Ο Καρλ Σλούτερ. Γεια σας. Ε, ε, ε, καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Θα... Ήθελα να συμφωνήσω μαζί σας όσον αφορά την υγεία και τον πλούτο. Είναι σημαντικός υπουργό Υγείας να μην εξετάζεται μόνο την καταπολέμηση των ασθενειών αλλά και την πρόληψη, τη διατήρηση της υγείας. Και είναι επίσης σημαντικό να βοηθήσετε και τον ε, Υπουργό Περιβάλλοντός σας, ε, τον Σάιμον, σε κάποιου από του αγώνε του, διότι αυτό βοηθάει ε, και τη δική σα οικονομία ε, ε, διατηρώντα την υγεία στου ανθρώπου. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να διατηρήσετε καλή ισορροπία στα θέματα αυτά. Είμαι υποψήφιο και ότι συζητήσε για την οδηγία για τον καπνό από την ομάδα των Πρασίνων. Έχουμε ένα πολύ Κάνω παράδειγμα από την Αυστραλία που θέλουν απλά πακέτα. Ε, ρωτήσανε ε, νέους ανθρώπους ε, αν θέλουν τσιγάρο προσφέροντάς τους από ένα απλό πακέτο από ένα πακέτο χωρίς τίποτα επάνω και διαπιστώθηκε ότι πράγματι ε, ε, λιγότεροι ζητούν τσιγάρο, αποδέχονται τσιγάρο δηλαδή όταν η συσκευασία είναι τόσο απλή. Έτσι λοιπόν αφαιρούμε ένα εργαλείο marketing από την ε, βιομηχανία. Άλλο θέμα που, με το οποίο θα ασχοληθείτε είναι οι κλινικέ δοκιμέ. Νομίζω ότι είναι σκανδαλώδε σήμερα ότι τα αρνητικά αποτελέσματα δεν δημοσιεύονται με τον ίδιο ρυθμό που δημοσιεύονται τα θετικά αποτελέσματα. Γιατροί συνήθως έχουν μόνο αποτελέσματα στα ε, δημοσιευμένα στοιχεία, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν ε, ε, λανθασμένες πληροφορίες οι γιατροί σχετικά με τις νέες θεραπείες. Δηλαδή, τα νέα φάρμακα δοκιμάζονται σε σύγκριση με το πλασέμπο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να δοκιμάζονται και με βάση την παλιά θεραπεία τα καινούρια, για να έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία και επίσης πολύ ανησυχητικό είναι ότι ο βασικός στόχος ε, στην ε, ε, στην κλινική δοκιμή είναι τα θετικά αποτελέσματα και εάν δεν φτάσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στον, στον βασικό στόχο του φαρμάκου αρχίζουν και ψάχνουν για δευτερεύουσες ε, ε, για, δευτερεύοντα αποτελέσματα. Για δευτερεύοντα αποτελέσματα. Ε, δηλαδή, αν δουν ότι δεν βοηθάει το φάρμακο σε αυτό που θέλανε, ε, προσπαθούν να βρουν κάτι άλλο στο οποίο να βοηθάει το φάρμακο αυτό. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, συνταγογραφούνται άχρηστα φάρμακα για άχρηστους ε, σκοπούς. Ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε να συνταγογραφούνται τα σωστά φάρμακα. Και επίσης ένας μηχανισμός που πιστεύω ότι θα πρέπει να δοκιμάσουμε στην Ευρώπη είναι... Πω πέρασαν ήδη τα τρία λεπτά. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των ε, τιμών ε, είναι ε, ένας νέος μηχανισμός που θα μπορέσει να μας βοηθήσει την παροχή φαρμάκων στις φτωχές χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μέσα σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όπως αναφέρθηκε είμαι εισηγητή για τον κανονισμό σε ό,τι αφορά τις διασυνορικές απειλέ, έχει ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος ή μάλλον θα ξεκινήσει μέσα στι επόμενες εβδομάδες και πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό κείμενο για το σύνολο των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών γιατί πράγματι πρέπει να προλαμβάνουμε και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις διασυνοριακές απειλές. Όπως είπατε, αυτό συνέβη και με τον ΙΤΑ 1 ή 1 ή με την γρήπη των πτηνών, αλλά και με το e Αν δείτε λοιπόν τι συνέβη τότε με το e αποδείχθη ότι αυτή η κρίση ε, προκλήθηκε και λόγω της ε, κακής επικοινωνίας και ότι η κακή επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ε, δυσμενείς επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές. Τώρα, για κάποια ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα ή ενδοκρινικοί διαταράκτες. Ε, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ε, χημικές ουσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ε, πολεμικής ανάμεσα στα θεσμικά όργανα που σχετίζονται βέβαια και με τον πόλεμο επιρροής ε, των βιομηχανικών κλάδων. Θα μας πείτε λοιπόν και μέσα στο επόμενο διάστημα τι ακριβώς θα να κάνετε από αυτού. Συμφωνώ με τη Φρανσάζ Γκοστέτ ε, ε, για το αλφακόλ που είναι ένα φάρμακο κατά των ε, σπάνιων ασθενειών κυρίως για τα νήπια και είναι τρομερό που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο φορές μάλιστα υπήρχε αρνητική γνωμοδότηση. Παρόλα αυτά, δόθηκε αδειοδότηση. Ενώ γνωρίζουμε ότι αυτό το φάρμακο ε, έχει και έναν ανταγωνιστή από τις ΕΠΑ. Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας ό,τι φορά την Ασπαρτάμι. Υπήρξε δημόσια διαβούλευση από την ΕΦΣΑ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί και εκεί είναι σημαντική διαμάχη σε ό,τι αφορά την Ασπαρτάμι και τις ε, συνέπειές της και εκεί είπατε ότι αν σήμερα ε, μας ζητούσαν να δώσουμε διοδότηση για να τεθεί στην αγορά ε, ο καπνός, δεν θα το κάναμε. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει τώρα και με, σε ό,τι αφορά την ασπαρτάμι. ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Υπουργό για την εξαιρετικά λεπτομερή ε, παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας. Με τα χαράς ε, βλέπω τον Υπουργό Υγείας της χώρας μου εντός της αιθούσης. Ελπίζω να βρείτε τα, τον τρόπο να συνεργαστείτε με τον κατάλληλο τρόπο με την Ιρλανδική Προεδρία. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, έχουμε ε, των, ε, τις οδηγίες για τον καπνό και για τον ιατρικό εξοπλισμό. Θα ήθελα να μπω κατευθείαν ε, στην ουσία και να σας θέσω ένα ζήτημα, ένα ερώτημα. Μιλήσατε για τις καινοτομίες, για την έρευνα. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο συζητούμε πολύ τη σημασία της πρόληψης και τη σημασία της ε, ύπαρξης ε, εκστρατιών ενημέρωσης και πρόληψης για τις, ε, για τις ασθένειες. Ήδη αναφέρθηκε το Health for Growth. Σε ό,τι αφορά την διεύρυνση, επέκταση κάποιων τομέων του προγράμματος, παράλληλα έχουμε ε, και τις ε, και ορισμένες ε, ασθένειες, τις εκφυλιστικές ασθένειες που είναι συγκεκριμένο και σημαντικό ζήτημα. E, Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, διάφορες ε, ασθένειες στις οποίες αναφερθήκατε, όπως επίσης και στον καπνό. Ε, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Ο πληθυσμός γυράσκει και η υγεία των ηλικιωμένων εξαρτάται από πολλά από αυτά που είπατε. Τα παιδιά μαθαίνουν ε, από τη συμπεριφορά των γονέων. Όταν το παιδί δεν βλέπει καλά παραδείγματα, τότε και σε μεγάλη ηλικία μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ε, κακή υγεία. Η εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί βάση για την πρόληψη των ασθενειών. Εάν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία μορφωμένη, τότε θα πρέπει ήδη σήμερα να ξεκινήσουμε τις προσπάθειές μας ε, και κατόπιν να φτάσουμε να μιλάμε για φαρμακολογία. Εάν δεν μπορέσουμε να συστηματοποιήσουμε τους βασικότερους τομείς, τότε στο μέλλον θα δούμε ασθένειες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ στις, στο Συμβούλιο να συνομιλήσετε με τους ε, ε, ομολόγους σας ε, σχετικά με την πρόληψη. Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο. Και επίση σε μια ασθένεια που υπάρχει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και αλλού είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη συχνά οφείλεται στον τρόπο ζωής. Θα πρέπει να προσέξουμε ε, ώστε να μην δούμε αύξηση το, της κατάθλιψης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Οκονή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβαλλοντικών Υποθέσεων. Ε, ε, ένα σημείο μόνο. Χθε διοργάνωσα μία συνδιάσκεψη με τον καθηγητή Βαλά, που είναι Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων. Μας ε, μίλησε εκτενώς ε, για τις ε, πανδημίες που προκαλούνται από τα ζώα. Το 60% των παθογενειών που πλήττουν τους ανθρώπους προκαλούνται από τα ζώα. Αυτή είναι η βασική τους προέλευση. Ποια είναι η σύνδεση λοιπόν, μεταξύ, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ αυτού του διεθνούς παρατηρητηρίου ε, που εκπροσωπεί 78 κράτη-μέλη ε, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι επαφές λοιπόν που υπάρχουν μεταξύ του Συμβουλίου και αυτό το Διεθνές ε, Παρατηρητήριο Ζωικής Υγείας και αν όχι, μήπως θα ήταν, αν δεν υπάρχουν τις επαφές, μήπως θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθούν. Γιατί έχουν εξαιρετικές πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα της υγείας των ζώων, των πανθογενειών ε, των πανδημιών και το καθεξής, αλλά και το γεγονός ότι και άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, ενδεχομένως να έχουν διάθεσή τους εξαιρετικές πληροφορίες και να μπορούν να συνεργαστούν και μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις ερωτήσεις. Θα τις πάρω με τη σειρά. Κυρία Μακέβεν, χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιλογή σας ως συγγήτρια για την έκθεση και ευχαριστώ για την υποστήριξη ώστε να προχωρήσει αυτή η οδηγία αν δεν εκφράσετε και εσείς αυτή την στοιχεία, μπορεί να μην τα καταφέρετε. θεωρείτε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για όλους για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών μας. Τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρατε για το άσθμα είναι πολύ καλά ουσιαστικά που μας δώσατε. Και παρά τα πολύ ψηλά ποσοστά καπνιστών που δεν δείχνουν πειθαρχία και δεν πιστεύουν σε αυτά τα στοιχεία, πάντως ε, η αλήθεια είναι ότι είναι ενθαρρυντικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το μονοξίδιο του άνθρακα, δεν είναι ακριβώς θέμα αρμοδιτάσμου, μου. Πράγματι όμως μπορεί να προκαλέσει τραγωδίες και πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου θα πρέπει να διαφημίσουμε, να κάνουμε εξαρτήσεις ενημέρωσης προς τους πολίτες για να καταλάβουν ε, τι κίνδυνος ολοχεύει από το μονοξείο του άνθρακα στο σπίτι. Αλλιώς καταλήγουμε σε τραγικές καταστάσεις. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τις κλινικές δοκιμές, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Ξέρετε, ως γιατρός, χαιρόμουν όταν έβλεπα ένα καινούργιο προϊόν να βγαίνει στην αγορά και έβλεπα ότι το 1 δέκατο του κόστους ε, ήταν το, η ενεργό ουσία. Και η ενεργό ουσία ήταν η ίδια. Ε, Αναρωτιόμουν λοιπόν γιατί θα πρέπει να στοχογραφήσω ένα νέο φάρμακο. Θα πρέπει να το γνωρίσουν αυτό οι γιατροί. Όταν στοιχογραφούν πολύ ακριβά φάρμακα, κάνουν κακό ε, το σύστημα υγείας της χώρας ε, που θα μπορούσε να ταπανίσει αυτά τα ποσά κάπου αλλού που είναι απόλυτα αναγκαία. Θα πρέπει λοιπόν ε, και τα φαρμακευτικά εργαστήρια, οι φαρμακευτικά εταιρείε, αλλά και οι γιατροί έχουν ένα καθήκον έναντι των ασθενών, αλλά όχι μόνο του συγκεκριμένου ασθενούς, αλλά έναντι όλων των ασθενών και του συμφέροντών τους. Βεβαίω η καινοτομία και η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει ε, να την παρακολουθούμε. Είναι ένα τομέα πολύ ε, ε, ενδιαφέρον να τον παρακολουθεί. Αλλά δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι το νέο και ακριβό φάρμακο είναι και το απόλυτα καλό για τον ασθενή. Για τον κύριο Πανίου και τις δυσμενειακές απειλές. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Το παρακολουθούμε και εργαζόμαστε σκληρά μαζί με την Κομισιόν και οι Κύπροι φίλοι μας έκαναν πολύ καλή δουλειά στον τομέα αυτό και εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε αυτή τη δουλειά. Μιλήστε για συγκεκριμένου ε, παράγοντες, ε, για τις αταραχές που προκαλεί το κλίμα και άλλες χημικές ουσίες. Ο συνάδελφός μου, ο Υπουργός Τζον ε, Μπρούκνερ, έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον στον τομέα αυτό και το παρακολουθεί. Αναφερθήκατε σε ένα φάρμακο, στάφακολ. Και επίσης αναφερθήκατε και στις γλυκαντικές ουσίες ε, στα ροφήματα είναι μια διαδικασία που την εξετάζουμε, μελετούμε το θέμα και θα δούμε πού θα μας οδηγήσει. Τώρα για την πρόληψη. Αυτό είναι θεμελιώδη σημασία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Το είπα και στο Συμβούλιο στο παρελθόν. Εμεί ω πολιτικοί πρέπει να το πούμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, είναι πολιτικά πιο δελεαστικό να γενιάζει κανείς ένα νέο νοσοκομείο, ένα νέο ακριβό ιατρικό μηχάνημα, παρά να γενιάζει μια νέα διαδικασία για την υγεία. Άρα και είμαστε και εμείς υπόλογοι. Από τα λόγια πρέπει να περάσουμε στα έργα. Η πρόληψη κοστίζει λεπτά αλλά πολύ λιγότερα λεφτά από τη θεραπεία. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που λέγαμε για το καπνό. Αυτό θα προστατεύσει την υγεία των παιδιών μας. Δεν θα εισπράξουμε όμως, αν θέλετε, εμεί αυτή την πολιτική επιτυχία, γιατί αυτό θα συμβεί πολύ μακριά χρονικά στον ορίζοντα. Το θέμα είναι αν είμαστε κι εμείς σοβαροί και κοιτάμε α, διορατικά το μέλλον και θέλουμε να ε, κάνουμε κάτι ουσιαστικό. Για την πρόληψη των ασθενειών, αυτό που είπατε συμφωνώ απόλυτα και μαζί με άλλους ε, αρμόδιους υπουργούς, όχι μόνο τους υπουργούς υγείας, υπουργούς περιβάλλοντος, παιδείας, δικαιοσύνης, πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι άνθρωποι και τα παιδιά μεγαλώνουν. Η πρώτη και βασική εκπαίδευση γίνεται στο σπίτι, Αν θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα, τους γονείς, καθώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει τα παιδιά σε πολλούς ε, τομείς. Το θέμα των ε, ψυχικών νοσημάτων, ε, κατάθλιψη κτλ. είναι ένα τομέα στον οποίο σίγουρα πρέπει να κάνουμε έρευνα, να επενδύσουμε. Ξέρετε, πολύ συχνά τα ψυχικά νοσήματα είναι στα χτωπούτα κάθε συστήματος υγείας και σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Σίγουρα ο τρόπος ζωής, το lifestyle, επηρεάζει πάρα πολύ όλα αυτά ε, τα πράγματα. Η σωματική άσκηση βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο να αισθάνεται, να νιώθει καλύτερα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Και σίγουρα ένα πράγμα δεν είναι η και για τα πάντα. Ε, ό,τι αφορά την πρόληψη και την ε, εκπαίδευση θέλω να σας πω ότι στο άτυπο ε, συμβούλιο που θα έχουμε το Μάρτιο στο Δουβλίνο θα εστιάσει ακριβώς τη ζητήματα στα θέματα εκπαίδευσης, παχυσαρκίας και κακών αν θέλετε συνηθιών ζωής και πώς επηρεάζουν την υγεία μακροπρόθεσμα. Σύγχρονες κοινωνίες, σύγχρονος τρόπος ζωής και πώς επηρεάζει αν θέλετε αυτό την υγεία. Ε, διατροφή με υψηλή πρόσληψη θετανθράκων ε, χαμηλή έως μηδαμινή σωματική άσκηση. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Άνθρωποι που έχουν μια ισορροπημένη διατροφή και δεν έχουν προβλήματα υγείας. Αν πολύ απλά τους εισάγουμε το ψωμί ε, και τη ζάχαρη στη διατροφή, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Λοιπόν, για το παρατηρητήριο και για το ρόλο του Συμβουλίου συμφωνώ και εγώ. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σα, γι' αυτό υπάρχει και το Συμβούλιο. Όταν υπάρχει μια καλή πρακτική πρέπει να διαδίδεται ειλικρινά πάντοτε όταν δεν καταφέρουμε κάτι καλό να το περνάμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας, αυτό με εκπλήσει αρνητικά, δεν το καταλαβαίνω πώς γίνεται. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα ερωτήματα που μου δώσατε. Να απαντήσω. Ευχαριστώ τον Υπουργό για τη συμμετοχή του και την απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Εύχομαι σας προσωπικά και στην Ελληνική Προεδρία καλή επιτυχία. Ό,τι καλύτερο για το επόμενο εξάμεινο. Είναι πολλά τα πράγματα που έχουν δρομολογηθεί και είναι εξέλιξη. Χρειάζεται νομοθεσία. Αλλά καλή στρατηγική. Ο τομέα υγεία είναι ένα καλό τομέα πολιτική που μπορεί κανεί να δείξει τα ωφέλη που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε όλου του πολίτε. Σα ευχαριστώ και πάλι. Καλή τύχη.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωράμε με το διάλειμμα. Θα τα ξαναπούμε στις 3 η ώρα. Σας παρακαλώ θυμηθείτε τις κάρτες ε, της ψηφοφορίας σας ε, για να ξεκινήσουμε αμέσω με τις ψηφοφορίες, ε, διότι έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Σας εύχομαι καλή όρεξη.